Jó napot kívánok, kedves képviselőtársaim! Megkérek mindenkit, hogy eh, Σας καλωσορίζω όλους θερμά. Σας παρακαλώ να καθίσετε για να αρχίσει η συνεδρίαση για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Σας καλωσορίζω θερμά και πάλι και σας παρακαλώ να λάβετε θέσεις για να συνεχιστούν οι ψηφοφορίες. Είμαστε στο σημείο 48 στην ημερήσια διάταξη. Ε, Γενικός Προϋπολογισμός της Ένωσης, Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τροπολογία παριθμών 1. Υπέρ. Επαναλαμβάνω. Είμαστε στο θέμα υπαριθμών 48 απαλλαγή για το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τροπολογία παριθμών 1. Ψήφι Κατά. Αποχές. Απορρίψετε. ψήφι του συνόλου της πρότασης για την απαλλαγή. Ζητώ συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος. Ηλεκτρονικά θα πρέπει να ψηφίσουμε την τελική ψηφοφορία. Άρχεται λοιπόν. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Mindenki szavazott. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται λοιπόν. Szavazására. Συνεχίζουμε. A Júri egyes számú módosítója. Η ένα της νομικής επιτροπής υπέρ κατά ε, αποχές εγκρίνεται. Οι δύο της νομικής επιτροπής υπέρ. Α, θέλετε να τις ψηφίσουμε όλες μαζί. από τη 2 μέχρι και την 7, unblock. Γιούρι 2 μέχρι και ε, Γιούρι 7. Αν συμφωνείτε, να τις ψηφίσουμε όλες μαζί. Είπε Κατά. από την τροπολογία 2 της Γιούρη μέχρι την 6 της Γιούρη, διορθώνει ο Πρόεδρος. Στην παράγραφο 5 είναι. az Λοιπόν, Ψήφι υπέρ. 2 με 6 της Γιούρη. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Τώρα θα ψηφίσουμε την τροπολογία 7 της Γιούρη υπέρ. Όχι, στην παράγραφο 16. Ψηφίζουμε την τροπολογία υπεριθμών 7, όχι της Γιούρη, συγγνώμη, του κύριου Έρενχάουζα. Ψήφι υπέρ. Είναι τελευταία τροπολογία στον κατάλογο. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα το σύνολο ηλεκτρονικά αρχίζει τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και συγχαρητήρια στον εισηγητή. Ερχόμαστε τώρα στο σημείο 49 της μέσης διαταξής. Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ελεγκτικό συνέδριο. Η τροπολογία υπαριθμών 1. Ψήφι Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά το σύνολο της απόφασης. Πέρας. Σοσιαλιστές και δημοκράτες είναι ένας υπεράριθμος. Ποιος ψηφίζει. Ο κύριος Γκάιερ. Έχουμε αρκετούς σοσιαλιστέ παρόντες. Θα ήθελα να κάνω μία πρόταση. Ε, λοιπόν, δεν ψηφίζω εγώ. Θα μπορούσα να σας πω ότι το πρωί είχαμε ένα λιγότερο, αλλά δεν πιστεύω να πιάσει αυτή η δήλωση, οπότε θα ψηφίζω εγώ. <laughs> Okay. Okay.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 Ζητώ συγγνώμη, λέει ο κύριο Μπράτμπορν. Έχω πρόβλημα, δεν ε, μεταφράζονται αυτά που λέτε στα αγγλικά. Υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Εγώ τι να σας κάνω τώρα. Ε? Να τα λέω αγγλικά. Τώρα είναι εντάξει. Ε, με τη διαρμηνία. Τα ελληνικά είναι εντάξει πάντως. Λοιπόν, ας το ξαναπροσπαθήσουμε. Έλεγα λοιπόν ε, να ψηφίσουμε αν συμφωνείτε Εντάξει τώρα, ακούτε και τα αγγλικά. Μπορούμε να προχωρήσουμε. Συμφωνείτε από την τροπολογία 2 μέχρι και τη 10 να τις ψηφίσουμε μαζί. Unblock. Δεν συμφωνείτε. Ποιος δεν φωνεί. Καλά. Ψηφίζουμε την τροπολογία υπαριθμών 2. Ψηφίπε. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία παριθμών 3. Περ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία παριθμών 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία υπέρ 5. Ψηφί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συνεχίζουμε. Έχουμε τώρα την τροπολογία παριθμών 7. Ψηφί περ. Συγγνώμη, διορθώνει ο πρόεδρος ξέχασα την 6. Τώρα θα ψηφίσουμε την 6. Ψήφιπε. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τώρα είμαστε στην 7. Όχι, ηλεκτρονική επαλήθευση για την 6. Παρακαλώ, ψηφίζουμε την τροπολογία παριθμών 6 και την ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Αν ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία επαρθών 7. Ψήφι περ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία επαρθών 8. Ψήφι περ κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία υπεριθμών είναι ναι. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία υπαριθμών όχι, τι θέλετε, έλεγχο για τη 10 παρακαλώ ε, την ενέα, συγγνώμη, ε, διορθώνει ο Πρόεδρος. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία υπερθμών 9 ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται. 12-es παραγραφούς συνεχιζουμε η τροπολογια υπερθμών Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι έχει εγκριθεί, αλλά για καλό και για κακό ας το ελέγξουμε παρακαλώ. Η ηλεκτρονική επαλήθευση στην παράγραφο 12 τροπολογία υπαρθμών 10. Αυτό ελέγχουμε. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 12α, η τροπολογία υπαρθμών 11 ψήφι, πέρα κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία υπαριθμών 12 ψήφιπέ κατά εγκρίνεται. Η τροπολογία υπαριθμών 13 ψήφιπέ κατά αποχές Εγκρίνεται. Η τροπολογία παρθμών 14 ψήφι Κατά. Αποχές. Απορρίφτεται. Λοιπόν, τώρα το σύνολο του ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Δεν κρίνεται. Συνεχίζουμε. Σημείο 50. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Πάντα για την απαλλαγή του 2011. Η τροπολογία υπαριθμών 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η πρόταση τώρα όπως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικά ψηφίζεται. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα, οι επόμενες τροπολογίες, υπαριθμό 3, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία υπαριθμό 4, υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται. 5-6 έχουν αποσυρθεί. Η τροπολογία υπαριθμών 7. Εδώ υπάρχει, λέει, μια προφορική τροπολογία από πλευρά των σοσιαλιστών και με αυτή την αλλαγή ψηφίζουμε. Ψήφι κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία υπερθυμών 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές Τι έγινε, κουραστήκατε από τώρα. Δεν έχω καταλάβει πάρα πολύ το αποτέλεσμα, γι' αυτό θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Την τροπολογία παριθμών 8. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 9. Υπέ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία παριθμών 10. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία παριθμών 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία παριθμών 12. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία βαστών 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συνεχίζουμε. Το πλογή παρελθόν 16 Πε. Κατά. Αποχές. Είναι πολύ μικρή διαφορά και δεν μπορώ να καταλάβω. Ας το ελέγξουμε. Ε, αρχίζει λοιπόν η ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία παρελθόν 16. Εγκρίνεται. Η τροπολογία υπάρχει 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι έχει εγκριθεί, αλλά στο ελέγξουμε για καλό και για κακό. Ηλεκτρονική επαλήθευση λοιπόν για την τροπολογία 18 αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Για του κύριου Σόνικ. Τροπολογία αυτή. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία παριθμών 19. Ψήφι Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία παριθμών 20 της κυρίας Αγιάλα Σέντερ. Με μια προφορική τροπολογία δίπλα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία παριθμών 21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία υπάρχει 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και το τέλος 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και τώρα το σύνολο του ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικά αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Σοβαζάστ Λεζάρουμ. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην Επιτροπή των Περιφερειών. Τροπολογία 1 ψήφι Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία τώρα για την απαλλαγή. Πέρας. Εγκρίνεται. πρόταση ψηφίσματος. Τροπολογία 2. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Υπέρ, κατά. Α, θα επιστρέψουμε στην 2. Ας κάνουμε λοιπόν ηλεκτρονική επαλήθευση για την υπαριθμόν 2 τροπολογία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τώρα, τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Υπαριθμόν 5 τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά Άποχες. Εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται αυτή. Τώρα το τροποποιημένο ψήφισμα η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Έκλεισε τέλος δηλαδή της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και Συνεχίζω με το θέμα 52. Ευρωπαίος συνήγορος του πολίτη, η διαμεσολαβητής. Πρώτη τροπολογία, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται για την απαλλαγή, ηλεκτρονική ψηφοφορία αρχίζει. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογίες για το ψήφισμα. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και αυτή. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παριθμόν 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία για την τροπολογία υπαριθμών 7. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και αυτή. 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τώρα η πρόταση ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικά αρχίζει η ψηφοφορία Τέλος. Εγκρίνεται. Τέλος. Τροπολογία, ε, συγγνώμη με συγχωρείτε, απαλλαγή του εντεταλμένου την προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι και το τελευταίο παράγραφος 1, τροπολογία 1, ψήφι υπέρ. Αυτά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία τώρα για την πρόταση αρχίζει πέρας εγκρίνεται. Προχωρώ στις τροπολογίες. Τροπολογία λίμπε, δηλαδή θεμελιωδών ελευθεριών, 2 υπέρ. Παραλαμβάνω, λίμπε 2. Τροπολογία 1, λέει ο τώρα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και αυτή. Παράγραφος 5. Τροπολογία του κυρίου Σόνικ. Υπαριθμών 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και αυτή. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τέλος. Τροπολογία 4 της Επιτροπής Θεμελιδών Ελευθεριών. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και αυτή. Και τώρα η ηλεκτρονική, δηλαδή ονομαστική ψηφοφορία για το τροποποιημένο ψήφισμα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Η πρόταση εγκρίθηκε. Για σήμερα λοιπόν εδώ ολοκληρώθηκε ο κύκλος των ψηφοφοριών. Σας ευχαριστώ όλες και όλους και συγχαίρω τους εισηγητές, καθώς επίσης και τις συνεργάτητες και τους συνεργάτες της Γραμματείας. Number 46. Yes, now is the study. Yes. Ο πρόεδρος συνεχίζει. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε με την ημερησία διάταξή μας στο επόμενο θέμα μελέτη για τις διαφορές στην δυτική απόδοση μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την ανάκτηση παραδοσιακών ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα γίνει παρουσίαση της μελέτης, θα ακολουθήσει συζήτηση. Το λόγο δίνω αμέσως στην κυρία Εστέρ Ντελάνγκε. Thank you. Uh, thank you very much, uh, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα το γυρίσω στα Ολλανδικά όμως για αλλαγή, διότι τώρα μπαίνουμε σε μια προβληματική που είναι αρκετά περίπλοκη από τη φύση της. Είναι η παραδοσιακή ήδη πόρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως γνωρίζετε είναι αυτό που θα πρέπει να κλείσει το προϋπολογισμό μας. Οι παραδοσιακοί ήδη πόροι ε, φύνουν και θα πρέπει να τα προσαρμόσουμε με εθνικές συνεισφορές. Δηλαδή όσο μικρότερη είναι παραδοσιακή ήδη πόρη και όσο λιγότερο ε, μειώνονται οι παρατυπίες και οι αδασταλίες, τόσο περισσότερο θα πρέπει να βάλουν και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό θα πρέπει να γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ε, τι γίνεται με τις ε, επιστροφές των αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών, ε, τι γίνεται με τους ιδίους πόρους και επειδή εμείς δεν ξέρουμε όλες τις λεπτομέρειες, δεν ξέρουμε ας πούμε τι γίνεται στο έκτο ψηφίο μετά την υποδιαστολή, γι' αυτό ζητήσαμε μια μελέτη, τι κάνουν τα κράτη-μέλη, ποια έχουν καλύτερες επιδόσεις, ποια λιγότερο καλές, για να μπορέσουμε να βγάλουμε τα συμπεράσματα και τα διδάγματά μας στην Επιτροπή Ελέγχου και από τις χώρες που, πώς να το πω, έχουν καλύτερες επιδόσεις, για να μπορέσουμε ε, να προσαρμοστούμε και οι υπόλοιποι. Ε, δεν θέλω να φάω εγώ πάρα πολύ χρόνο. Αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο ζητήσαμε αυτή τη μελέτη και κάναμε αυτή την ανάθεση και τώρα νομίζω ε, θα μπορέσουμε να περάσουμε, να δώσουμε το λόγο σε εκείνους που έκαναν τη μελέτη, να μας την παρουσιάσουν και να δούμε ποια είναι τα ευρήματά τους από αυτών των θεμάτων. Αυτά τα ολίγα και σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ τους ε, κυρίους που θα μας παρουσιάσουν την μελέτη να λάβουν το λόγο. Ε, Παρακαλώ ανοίξτε το μικρόφωνο για να σας ακούσουμε και να προχωρήσουμε. Λοιπόν, ονομάζομαι James Spencer, ε, είμαι Ονομάζομαι James Πένς, είμαι συνταξιούχο αξιωματούχο Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή τη στιγμή διδάσκω πολιτικέ επιστήμε στο Παρίσι. Ε, μαζί μου θα είναι και ο, ο συνάδελφο Hans Davids τη Your Balance Αυτό θα ξεκινήσει. Λέγομαι Hans Davids. Ε, είμαι παλαιός υπάλληλος ε, τη της εφορίας κάτω χώρες. Ε, και πρέπει να σας πω ότι έχω δουλέψει και στην διαχείριση και διοίκηση των τελωνίων. Ε, δούλεψα 8 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού και στην Όλαφ ε, και συγκεκριμένα εργάστηκα την ανάκτηση παραδοσιακών ίδιων πόρων ενώ στην Όλαφ ασχολήθηκα με τις παραβάσεις και τις ατασταλίες. Ε, ξεκίνησα πριν από λίγο καιρό μια εμπορική ε, διαδικασία έτσι ώστε να διευκολύνουν τις χώρες μέλη στην ανάκτηση των παραδοσιακών ιδίων πόρων τους. Ε, ξέρουμε πια ε, πώς, από τι αποτελείται ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ σας δίνω ένα παράδειγμα ε, του 2011, του προϋπολογισμού του 2001 έχουμε εδώ τις εισφορές των κρατών, τις εθνικές εισφορές 68%. βλέπουμε το ΦΠΑ που είναι το 11%. Βλέπουμε την ανάκτηση των παραδοσιακών ιδιοπόρων και βλέπουμε βεβαίως και το πλεόνασμα από τα προηγούμενα ε, έτη ε, τα οποία λαμβάνονται υπόψη. Ε, τα έσοδα πρέπει να είναι ισοσκελισμένα με τις δαπάνες και γι' αυτό ακριβώς οι ίδιοι πόροι παίζουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ε, μια και η εθνική συνεισφορά είναι το εξισορροπητικό ε, στοιχείο, είναι πολύ σημαντικό να καθορίσουμε ε, αυτό το, το τμήμα του προϋπολογισμού και επίσης είναι σαφές σύμφωνα με αυτό το σχήμα ότι εάν κάποιες χώρες δεν μπορέσουν να ανακτήσουν τους παραδοσιακούς είδους πόρους τότε θα πρέπει να αυξήσουν την εθνική τους συνεισφορά. Ε, αυτή η μελέτη έχει χρησιμοποιήσει στο μέτρο του δυνατού ε, στοιχεία τα οποία είναι δημοσιευμένα, τα οποία επίσης είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό, καθώς επίσης ε, και τις δημοσιεύσεις της Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης. και τα στατιστικά παραρτήματα, καθώς επίσης ε, τους ετήσιους λογαριασμούς και την ετήσια έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Προϋπολογισμού. Έχουμε εδώ παραθέσει ε, και την ε, κατάτμιση ανάλογα με τις εισφορές των κρατών μελών ε, υπογεγραμμένους από το Κολέγιο των Επιτρόπων για να έχετε και μια καλύτερη ιδέα σύμφωνα με τις συνθήκες ε, απαιτείται προς το οικονομικό συμφέρον, ε, μάλλον απαιτεί το οικονομικό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να διαφυλαχθεί. Και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μια διαδικασία ταυτοποίησης των παρατυπιών και των ατασταλιών μέσω και νομικών διαδικασιών, ακόμα και ενώπιον των δικαστηρίων και αυτό έχει καλά αποτελέσματα. Τα κράτη-μέλη και τα τελωνία τους ε, διαφέρουν μεταξύ τους και όσον αφορά την οργάνωση και όσον αφορά τις νομικές αρμοδιότητες και εξουσίες και όσον αφορά τις διευρυμένες αρμοδιότητες που μπορεί να έχουν. χρησιμοποιώντας πάντα στοιχεία τα οποία είναι ε, δημόσια διαθέσιμα όσον αφορά την, ε, τον ποσό, το ποσό ανάκτησης ε, από τα τελωνία στα κράτη-μέλη, βλέπουμε μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας αυτής, που εφ' εξής θα ονομάζομαι απόδοση ή μάλλον επίδοση των κρατών μελών. Το ερώτημα που προκύπτει λοιπόν είναι το εξής. Ε, ποια είναι η διαδικασία ανάκτησης παραδοσιακών ε, ιδίων πόρων. Ε, έχουμε εμεί ταυτοποιήσει πέντε διαφορετικά σημεία ή έτσι, φάσεις της διοικητικής διαδικασίας. Δεν υπάρχει μαύρη μαγεία εδώ, είναι όλα πάρα πολύ απλά. Αυτά τα πέντε πεδία λοιπόν ε, είναι ο έλεγχος, ε, η προσπάθεια ταυτοποίησης των παρατυπιών, ε, η προσπάθεια καθορισμού ενός μια στάνταρ διαδικασίας για τα τελωνία και βεβαίως και μέσω των ελέγχων ροή χρημάτων προς τις Βρυξέλλες το σύστημα είναι σαν να έχει μόνο είσοδο και όχι έξοδο με την έννοια ότι από τη στιγμή που μπαίνεις στο σύστημα περνάς από τα διάφορα στάδια ε, και ε, σε κάθε στάδιο θα πρέπει ε, να δείξεις μια συγκεκριμένη επίδοση. Εάν μπει κανεί λοιπόν στη διαδικασία αυτή πρέπει να περάσει από αυτά τα πέντε βήματα πριν ε, στείλει χρήματα στι ε, Βρυξέλλες. Σημαίνει επίσης ότι εάν ένα από αυτά τα βήματα αποτελεί τον ασθενή κρίκο τότε θα έρθουν λιγότερα χρήματα. Επίσης σημαίνει ότι όταν κανείς ε, είναι σε θέση να συνδυάσει αυτά τα πέντε ε, στάδια σωστά, μπορεί να φέρει πολλά χρήματα και επομένω περισσότερους παραδοσιακούς ίδιους πόρους στις Βρυξέλλες. Θα καταλάβατε, ε, φαντάζομαι, ότι σε όλα αυτά τα στοιχεία μπορεί κανείς ε, να ε, διαπιστώσει ότι όσο πιο σαφή ε, υλοποίηση έχει το κάθε από αυτά τα πέντε βήματα, τόσο πιο καλό είναι το αποτέλεσμα. Και εάν προσθεθούν αυτά τα πέντε βήματα, τότε μπορεί κανείς να βρει το σύνολο των παραδοσιακών ίδιων πόρων που τελικά θα φτάσει στις Βρυξέλλες. Βεβαίως ότι ισχύει για την καλή επίδοση, ισχύει και για την κακή. Το αντίθετό του μάλλον ισχύει για την κακή. Όταν μιλάμε ε, για επίδοση ε, ε, είναι κάτι θετικό, το αντίθετό του είναι η διάχυση ε, και βεβαίως ε, όλα αυτά τα χρήματα τα οποία περνούν από αυτή τη δεύτερη διαδικασία δεν φτάνουν ποτέ στις Βρυξέλλες. Είναι ενδιαφέρον να δει κανεί σε ποια σημεία των κρατών μελών, σε ποια σημεία της διοίκησης ή των τελωνίων εξαερίζονται αυτά τα, εξανεμίζονται αυτά τα χρήματα. Ε, μία μελέτη λοιπόν των στοιχείων αυτής της διαδικασίας απώλειας των ε, πόρων θα μας ε, δώσει να καταλάβουμε πώς έχει η διαδικασία. Αμοιβαία αναγνώριση των ε, διαφόρων στοιχείων, συσχετισμός ανάμεσα στα θετικά και τα αρνητικά μπορούν τελικά να μας δώσουν στο καταληκτικό συμπέρασμα σχετικά με το τι συμβαίνει στα τελωνία. Αυτό που είναι καινούριο στην προσέγγιση μας είναι ότι σε κάθε στάδιο της διπλής αυτής διαδικασίας, είτε δηλαδή της ε, απόδοσης, ε, είτε της ε, εξαφάνισης κατά κάποιο τρόπο των χρημάτων, μπορέσαμε να μελετήσουμε λέω, το κάθε, την, το, την κάθε μεμονωμένη διάδα και κατά κάποιο τρόπο να βρούμε και, μία, και ένα σκορ και μία επίδοση, όχι μονάχα για τα μεμονωμένα βήματα, αλλά και για το σύνολο και το κάναμε για αυτό για όλες τις χώρες μέλη και για μια εξαετή περίοδο. Επομένως ε, η άσκηση αυτή ήταν πολυετής, ε, αφορούσε πολλά κράτη-μέλη και αφορούσε και πολλά στάδια. Το σύνολο των στοιχείων μας ε, έδωσε πολύ αξιόλογα, πολύτιμα μπορώ να πω, στοιχεία. Όπως θα έχετε διαβάσει ήδη στην έκθεση, για κάθε μία από τις μεμονωμένες χώρες είμαστε σε θέση να βρούμε ε, πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Πρώτα απ' όλα, διαπιστώσαμε διαφορές. Διαπιστώσαμε μάλιστα ουσιώδεις διαφορές. Και μάλιστα, εάν δει κανείς ε, ε, υποπροπτική αυτά τα έξι χρόνια, διαπιστώσαμε ότι οι διαφορές είναι διαρθρωτικές, ακολουθούν ένα συγκεκριμένο στυλ και, μια συγκεκριμένη, και έχουν μια συγκεκριμένη μορφή. Ε, συνδυάζοντας τους βαθμούς επίδοσης στο σύνολο των ανακτηθέντων παραδοσιακών πόρων, είμαστε σε θέση εν τέλει να κάνουμε και κάποια εκτίμηση για το ύψος των χρημάτων και γι' αυτό καταλήξαμε λοιπόν στο, στο αποτέλεσμα ότι αν δει κανεί όλα τα κράτη-μέλη ε, σε, σε αυτές τις πέντε φάσεις για έξι χρόνια και αν όλα τα κράτη είχαν ε, την καλύτερη δυνατή επίδοση, τότε ενδεχομένως θα υπήρχε ένα ανακτηθέν ποσό το οποίο θα κυμαίνεται μεταξύ ε, ενός και τριών δις ευρώ για αυτήν την εξαετή περίοδο. Αυτό που ε, το συμπέρασμα που καταλήξαμε επίσης είναι ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, η επίδοση των τελωνίων ε, για την υποέρευνα περίοδο ήταν 0,7%. Θα αναρωτηθείτε τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι τα αποτελέσματα ανάκτησης όλων των ανιχνευθυσών παρατυπιών για ε, εκατοντάδες περιπτώσεις ε, που ηλέχθησαν ε, είναι περίπου 70 cents. Ίσως φαντάζεστε ότι με αυτό είναι πολύ λίγο. Αλλά όμως με τα χρόνια μάθαμε να χρησιμοποιούμε την εκτίμηση του 2% και θα δείτε, θα δείτε και αργότερα θα σας το δείξω ότι ε, ακολουθεί πτωτική πορεία ε, αυτή η διαδικασία. Αλλά ε, εάν χρησιμοποιήσουμε σαν δείκτη το 0,7% μπορούμε να συγκρίνουμε χώρες μέλη οι οποίες δεν μπορούν να συγκριθούν μεταξύ τους με την έννοια ότι έχουμε βρει μεταξύ αυτών των χωρών πάρα πολύ μεγάλες διαφορές. σε μερικές περιπτώσεις ε, οι διαφορές ανάμεσα στο καλύτερο αποτέλεσμα και το ε, χειρότερο αποτέλεσμα μεταξύ των κρατών μελών, ε, η σχέση, ο λόγος μπορεί να είναι 20 προς 1. Αλλά βεβαίως εδώ αναφέρομαι σε πολύ ειδικέ καταστάσεις, σε ειδικά κράτη-μέλη και σε ειδική χρονική στιγμή. Επομένως, ε, για τα πέντε στάδια που σας έδειξα προηγουμένως, ε, χρησιμοποιήσαμε πολύ συντηρητικές ε, εκτιμήσεις και βγάλαμε επομένως τις εκτιμήσεις που κάναμε την χώρα που βρισκόταν πρώτη στον κατάλογο και τη χώρα αντίστοιχα που βρισκόταν τελευταία στον κατάλογο. Επομένως, ε, εάν βγάλουμε και αυτές τις χώρες, ο λόγος ο οποίος παραμένει είναι 10 προς 1, δηλαδή εξακολουθεί η σχέση να είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τώρα θα ήθελα να σας ε, δείξω έναν πίνακα ο οποίος σας δίνει τα συνολικά αποτελέσματα στο τέλος της ε, εξαετούς διαδικασίας ε, και μάλιστα για τα πέντε στάδια της επίδοσης ε, που ανέφερα προηγουμένως. Αριστερά στο γράφημα βλέπετε το EU. Δηλαδή, αν πάρετε τους μέσους όρους όλων των κρατών μελών και τους βάλετε μαζί και, και, πάρετε ε, αυτό το αποτέλεσμα σαν ε, δείκτη μέσου όρου, τότε μπορείτε να συγκρίνετε τις επιδόσεις των κρατών μελών σε σχέση με αυτό το δίκτυ. Βεβαίως πρέπει να παραδεχτούμε ότι ένας τέτοιος δείκτης ε, είναι το αποτέλεσμα στατιστικής διαδικασίας και δεν έχει πραγματική ιδεοντολογική αξία Παρά τα αυτά όμως ε, μας βοηθάει έτσι ώστε να δούμε καθαρότερα την εικόνα αυτή. Γιατί διαπιστώνουμε ότι η διαφορά ανάμεσα στους πρώτους και τις τελευταίους ε, ή αν θέλετε καλύτερα την ψηλότερη επίδοση μείον ένα και τη χαμηλότερη μείον ένα ε, και μάλιστα σε μια εξαετή περίοδο είναι όχι μόνο μεγάλη αλλά και δείχνει διαρθρωτικές διαφορές. Κάτι άλλο που μας εκπλήσει νομίζω σε αυτό το γράφημα και που ε, μας έχει καταπλήξει σε, όλες τις, όλα τα γραφήματα που αφορούν τις επιδόσεις των κρατών είναι το εξής. Δεν είναι δύσκολο να κάνει κανείς διαφοροποίηση ανάμεσα στους υψηλούς, τους χαμηλούς και τους μέσους ε, σε, όρια, σε, όρους ε, επίδοσης. Και Ε, είδαμε ότι ο μέσος όρος κινείται σε ένα συν πλην 30% ενώ οι υψηλές επιδόσεις ξεπερνούν το 30% ενώ οι χαμηλές επιδόσεις ε, είναι σαφώς κάτω από το 30%. χρησιμοποιούμε το high και low performance, υψηλή και χαμηλή επίδοση στην έκθεσή μας, ε, έτσι ώστε να γίνει κατανοητή η, το, να γίνει κατανοητό το συμπέρασμα που προκύπτει από το γράφημα αυτό. Δεν θέλουμε με κανέναν τρόπο να ταξινομήσουμε τα κράτη-μέλη, απλώς καταδεικνύονται οι διαφορές όσον αφορά την ανάκτηση παραδοσιακών ιδίων πόρων μεταξύ κρατών μελών. Ήδη είπε ο συνάδελφος ότι οι υπηρεσίες της Κομισιόν στην συνήθη τους εργασία προσπαθούν ε, να ε, εξισορροπήσουν ή να εξουδετερώσουν αν θέλετε ε, τα προβλήματα και τις ελλείψεις στην ανάκτηση παραδοσιακών ιδίων πόρων. Αυτό που μας δείχνει τούτο το γράφημα είναι ότι κάτι τέτοιο, δηλαδή αυτό που προσπαθεί να κάνει η Επιτροπή ίσως δεν αρκεί. Διότι αυτές οι διαφορές μπορούν να μεταφραστούν σε χρήματα και τότε οι διαφορές μετριούνται σε εκατομμύρια. Το καθαρό δίδαγμα αυτής της εικόνας, ειδωμένο σε μια εξαετή περίοδο, μπορεί να φτάσει σε 2 μέχρι 4 δις, εκατο... δις ευρώ, λέω. Δηλαδή, είναι η διαφορά των χρημάτων που θα είχαν ανακτήσει τα τελωνία εάν είχαν ε, όλα λειτουργήσει βάσει της υψηλότερης ε, επίδοσης. Και εάν υπολογίσουμε ότι ήδη μιλάμε για μια διαφορά ενός δίσε, εάν ε, είχαν όλοι παραμείνει περίπου στον μέσο όρο, ε, τα επιπλέον χρήματα που θα είχαν ανακτήσει τα τελωνία θα ήταν ένα με τρία δις. Θα σας δείξω και κάτι άλλο. Εάν συμφωνήσετε με την παραδοχή μας ότι αυτό το ποσό των τριών δις ε, είναι το ε, μεγαλύτερο ποσό ε, ιδίων πόρων που θα μπορούσε να είχε ανακτηθεί, τότε το ερώτημα που προκύπτει λογικά είναι ποιος πληρώνει για αυτή τη διαφορά. Όσοι έχετε διαβάσει την έκθεση ε, θα έχετε διαπιστώσει ότι δεν έχουμε κάνει σχόλια επ' αυτού, αλλά ε, απλώς χρησιμοποιήσαμε τα γραφήματα έτσι ώστε να γίνει κατανοητή αυτή η διαφορά και σε εσά. Εάν όλα τα κράτη-μέλη είχαν εργαστεί όπως ας πούμε εργάζονται τώρα, τότε αυτά τα χρήματα θα είχαν πληρωθεί από τα κράτη-μέλη σύμφωνα με αυτό το γράφημα. Αυτό ας πούμε θα σήμαινε ότι η Γερμανία θα έπρεπε να πληρώσει περίπου μισό δις. Και γιατί αυτό? Διότι όπως βλέπετε σε αυτήν την εικόνα ε, υπάρχει η απώλεια των πόρων κατανεμημένη ανακράτος μέλος σύμφωνα με την ε, ε, έλλειψη παραδοσιακών ε, ίδιων πόρων. Και είναι η Γερμανία αυτή η οποία πληρώνει μια εισφορά της τάξης του 20%. Και επομένως με αυτό το 20% με το ίδιο ποσοστό συμβάλλει και στις απώλειε. Μπορεί κανείς να ρωτήσει ή να αναρωτηθεί κατά κάποιο τρόπο μήπως πρέπει να τιμωρηθεί ας πούμε η υψηλή ε, επίδοση σε σχέση με τη χαμηλή επίδοση ε, και ούτε αυτό το γράφουμε στην έκθεσή μας αλλά το δείχνουμε με το επόμενο γράφημα έτσι ώστε να καταλάβετε καλύτερα την κατάσταση. Έχουμε ε, την ε, εισφορά κατά κεφαλή ανακράτος και το αποτέλεσμα ανα ε, πολίτη, ανα ε, ψηφοφόρο, ανα ε, φορολογούμενο, η διαφορά λέω γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Εάν έχετε ψηλό GNI και χαμηλό πληθυσμό, τότε πληρώνετε πληρώνεται πολύ περισσότερο από ότι μία χώρα με υψηλό με υψηλό ΑΕΠ αλλά και υψηλό ε, κατά εισόδημα. Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με του υπολογισμού μα, ότι πληρώνει περισσότερο ο μεμονωμένο πολίτη του Λουξεμβούργου από ότι ο μεμονωμένο πολίτη τη Βουλγαρία. Και βεβαίω καταλήγουμε στο ίδιο ε, ε, συμπέρασμα ότι κάποιο πρέπει να πληρώσει για αυτά τα μη ανακτηθέντα παραδοσιακά ποσά, από του παραδοσιακού ίδιου πόρου δηλαδή. Και φτάνουμε λοιπόν σε δύο πίνακες τους οποίους θέλουμε να συγκρίνουμε. Ε, στον πρώτο πίνακα είναι, ε, βλέπουμε ένα πίνακα που τον είδαμε ε, και πρωτήτερα σε μια άλλη διαφάνεια. Δείχνει τα αποτελέσματα της συνολικής επίδοσης των τελωνίων την, τελευταία, την υποέρευνα εξαετία 2006-2011. Στο από κάτω γράφημα βλέπετε τους μεγαλύτερους εισφορείς με βάση το ΑΕΠ. Τώρα έχουμε και κάποια κόκκινα κράτη-μέλη, δεν ξέρω αν τα βλέπετε. Είναι οι καθαροί εισφορεί, οι οποίοι ταυτόχρονα όμως είναι και οι καλύτεροι μαθητές, αυτοί που έχουν την καλύτερη επίδοση σύμφωνα με, τις, ε, με τη δικιά μας μελέτη. Ε, κάνοντας τους αντίστοιχους υπολογισμούς ε, θα καταλάβετε ότι ότι περίπου χώρε μέλη, που είναι μεγάλη εισφορής είναι υπεύθυνη και για το 70% ε, των εθνικών εισφορών, αλλά έχουν και την υψηλότερη επίδοση. Μπορείτε επίσης να διαπιστώσετε ότι πολλά χρήματα θα μπορούσαμε να κερδίσουμε από αυτούς που δεν έχουν μεγάλη επίδοση και που δεν έχουν και μεγάλη ε, συνεισφορά. Σας δείχνουμε λοιπόν το καθαρό αποτέλεσμα εάν, ε, εάν συνεχίσουμε να μην ε, ενδιαφερόμαστε για την ανάκτηση των πόρων μέσω των τελωνίων. Ε, νομίζω ότι η εικόνα αυτή δείχνει σαφώς ότι πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα διαβάσω όλες τις συστάσεις και τα συμπεράσματά μας. Επιτρέψτε μου να σας πω λίγα μόνο για να σας εξηγήσω το πρόβλημα. Και πρώτο, ότι η Κομισιόν έχει δίκιο που προχωρεί και θεωρεί υπεύθυνα τα κράτη-μέλη, οικονομικά δηλαδή, για ζημιέ που παθαίνει ο κοινοτικό προπολογισμό, όταν μπορούν να εντοπιστούν. Εδώ βέβαια υπάρχουν δύο θέματα. Πρώτο σκέλος. Το δεύτερο σκέλος είναι η χρήση των στατιστικών με τακτικό τρόπο, όπως προτείνουμε και εμείς εδώ, και να εκμεταλλευτούν όλες τις ευκαιρίε για να αυξηθεί η συνολική οικονομική απόδοση της Ένωσης. μπορούν να αναλυθούν δράσεις με στόχο την βελτίωση της απόδοσης της διαδικασίας αυτής. Αν και δέχομαι ότι τα ποσά για τα οποία μιλούμε φαίνονται να είναι σχετικά μικρά όταν συγκριθούν με κάποια άλλα ποσά. Εάν δηλαδή βελτιώσει κανείς την ερμηνεία και πρακτική των στατιστικών των εθνικών λογαριασμών, τότε ίσως προκύψουν μεγαλύτερες εξοικονομήσεις από τον πόρο του ΑΕΠ. Και ανεξάρτητα, στην ουσία, από τις προτάσεις που κάνουμε εμείς εδώ. Οι χώρες μέλη πρέπει βέβαια να προχωρήσουν σε πραγματικά αυστηρή επανεξέταση του τρόπου με, τον οποίο συλλέγουν τους πόρους, τα δεδομένα να είναι πιο επιμελής, πιο έγκαιρες να γίνονται οι μεταφορές προς την Ένωση και να προχωρούν σε κριτική αξιολόγηση των δικών τους τελωνιακών συστημάτων. Εγώ είδα ότι το σχέδιο απαλλαγής αναφέρει τις δυσκολίες και σημείωσα ακόμη ότι ορισμένε από τις κριτικές παρατηρήσεις που γίνονται από το ελεγκτικό συνέδριο στην ετήσια έκθεσή του του 2011 όπου συζητούν το θέμα της απόδοσης των συστημάτων συλλογής των ιδιών πόρων τα επισήμανα αυτά λοιπόν παρακαλώ σκεφτείτε τις συστάσεις που κάνουμε και ελπίζω θα μπορέσετε να θεωρήσετε ορισμένε μπορείτε να τι εφαρμόσετε και στο μέλλον. Υπάρχουν και άλλες διαφάνειες που σας έχουμε παράσχει, που εικονογραφούν τα θέματα τα οποία έχουμε επισημάνει. Και θα μπορέσουμε να σας παραπέμψουμε σε αυτές την επόμενη συζήτηση. Σας ευχαριστώ κύριοι, κύριοι Σπέντς και Ντέιβις για την παρουσίαση των πολύτιμων αυτών σκέψεών σας. Ίσως η κυρία Εστέρ Τελάνγκε επιθυμεί να προβήσει κάποια σχόλια. Έχετε το λόγο. Ναι. Θα ήθελα να ακούσω βέβαια και την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν καταλαβαίνω καλά την έκθεση αυτή και είναι και πάρα πολύ τεχνικό το θέμα, τι λέγει, ότι τα κράτη-μέλη έχουν τόσο τεράστιες διαφορές που τη στιγμή που κάθε κράτος μέλος έχει κάποια επίδοση, ας πούμε αν ήταν όλοι στο επίπεδο του καλύτερου κράτους, αυτό τι σημαίνει ένα με δις για την περίοδο αυτή, δηλαδή 500 εκατομμύρια το χρόνο, αν θεωρήσουμε το ανώτατο όριο τρία δις που είναι ένα σχετικά μικρό κλάσμα ε, οι διπόροι παραδοσιακοί, αλλά είναι πολύ μεγάλη διαφορά στις επιδόσεις και στην απόδοση των κρατών μελών και μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδέχεται αυτές τις διαφορές μεταξύ κρατών μελών. Ε, σου λέει τι να κάνουμε, ε, κάθε χώρα έχει διαφορετική επίδοση, ενδεχομένω διαφορετική αντιμετώπιση και το βλέπω και συχνά αυτό να συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σου λέει ότι εντάξει είναι ευρωπαϊκοί οι κανόνες, όχι μόνο για τον προπολογισμό και σε άλλα επίπεδα, ξέρω εγώ από κάτι περιβαλλοντική νομοθεσία. Οι κανόνες είναι ε, ευρωπαϊκή, αλλά η έλεγχη τι να κάνουμε είναι εθνικό ζήτημα και υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην απόδοση, αλλά ναι, τι κρίμα, αλλά συμβαίνει αυτό και τι να κάνουμε. Θεωρητικά λοιπόν πιστεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι κάποια στιγμή θα ανακτηθούν αυτά τα ποσά, αλλά η ε, εμπειρία μας λέει ότι και 12 χρόνια μπορεί να περάσουν μέχρι να ανακτηθούν τα ποσά, αν ποτέ ανακτηθούν. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα και πάνω κάτω Αυτό που μας ενδιαφέρει για την απαλλαγή ως Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού είναι το εξής. Πώς θα αναλάβει και ποια πρωτοβουλία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να φροντίσει ακριβώς ε, χώρες να προσανατολίζονται προς τις καλύτερες επιδόσεις. Αντί να αφήσουμε αυτή την ψαλίδα να υπάρχει και να συνεχίζεται. Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι θα κάνετε το δέχεστε τυφλή σώμαση ότι τι να κάνουμε, εντάξει υπάρχουν διαφορές. Ελπίζω όχι. Γιατί πρόκειται για πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και δεύτερη ερώτηση, θέλω να ρωτήσω κάτι τους επιρρογνώμονες που έκαναν τη μελέτη. Αυτή η μεθοδολογία για την ανάκτηση ε, χρημάτων παίζεται σε πολλά γήπεδα. Ας πούμε στα διαρθρωτικά ταμεία, αλλά όχι μόνο. Αυτή τη μεθοδολογία θα τη χρησιμοποιήσετε και για τις εθνικές επιδόσεις στα διαρθρωτικά ταμεία, παράδειγμα. Δηλαδή, θα μελετήσετε και εκεί τι γίνεται. Γιατί με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα αυτό. Και πάλι αυτό που δεν με ενδιαφέρει εμένα είναι τι κάνει κάθε χώρα μεμονωμένα. Εντάξει, ενδιαφέρον είναι να το ακούμε και ως Ολλανδέζα ακόμα περισσότερο με ενδιαφέρει ε, γιατί έχουμε και εθνικό πρόβλημα, υπολοιπόμεθα τα τελευταία χρόνια και καλούμεθα να το βελτιώσουμε. Αλλά το θέμα είναι τι κάνει η Ευρώπη συνολικά για το μέλλον και πώς θα προχωρήσουμε. Δεν μπορώ εγώ να εξηγώ στους ε, πολίτες της χώρας μου ότι σε αυτούς τους τομείς χάνουμε 3 δισεκατομμύρια. Για τους ιδίους πόρους και μόνο, έτσι. Σε άλλους τομείς πολιτικής μπορεί να είναι ακόμα περισσότερα τα χρήματα. Δεν είναι καθόλου εύκολα αυτά και θα πρέπει να κάνουν βήματα και το λέω και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βελτιωθεί η κατάσταση. Πρώτον, τι θα κάνει η Επιτροπή για να τα βελτιώσει αυτά και δεύτερον, και προς ε, τους συντάκτες της μελέτης. Αυτή τη μεθοδολογία μπορούμε να την ε, ακολουθήσουμε και σε άλλους τομείς με shared management που έχει συνδιαχείριση και συνυπευθυνότητα το κράτος μέλος. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ελπίζω να μπορέσουν να απαντηθούν τα ερωτήματα αυτά της συναδέλφου. Καλωσορίζω θερμά τον κύριο Σόρτη, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του δίνω το λόγο. Είναι από τη Γενική Διεύθυνση Προπολογισμού. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή ε, που ζήτησε την έκθεση αυτή, την έρευνα αυτή, την οποία βεβαίως εμείς έχουμε διαβάσει. Άκουσα κάποια ερωτήματα προς την Επιτροπή, αλλά εγώ θα ήθελα να πω πρώτα απ' όλα ποια είναι η δικιά μας ανάλυση της έκθεσης αυτής, εάν μου επιτρέπετε. να πω ότι βεβαίως αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές ε, επιδόσεις ε, ανακράτη, μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά ε, την ανάκτηση των πόρων και βεβαίως και παρατυπίες οι οποίες ελέγχονται και από τις εθνικές διαδικασίες. Όμως τα ζητήματα αυτά δεν θα πρέπει να υπερεκτιμηθούν και θα πρέπει πάει πάση περιπτώσει να βγουν στις, σωστέ, στις σωστές τους διαστάσεις. 99 ε, φορές τις 100 ε, τα χρήματα τα οποία ανακτούν ε, οι χώρες με τον τρόπο αυτό μπαίνουν απευθείας στους ίδιους πόρους και βεβαίως υπάρχει το ποσοστό των παρατυπιών που όμως είναι μικρό και που εν τέλει ακόμα και μετά το τέλος των παρατυπιών ανακτώνται οι πόροι. Είδαμε στην, στα πλαίσια της έρευνας αυτής ε, και κάποια σχήματα, κάποια patterns τα οποία γνωρίζει ήδη ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα μελετά ε, η ερευνητική της μονάδα. Θεωρούμε βεβαίως ότι εδώ η προσέγγιση είναι πολύ στατιστική και πολύ θεωρητική και βασίζεται στην global analysis, στην συνολική ανάλυση. και ε, κυρίως ε, δείχνει το δάχτυ με το δάχτυλο τις χώρες οι οποίες έχουν χαμηλότερες επιπτώσεις. Από την άλλη πλευρά φυσικά ε, έχουμε και κάποιες δικές μας μελέτες από τις οποίες προκύπτουν κάποια στοιχεία. Ε, ας πούμε γίνεται λόγος στο ποσοστό ανείχνευσης των ε, παρατυπιών. Ε, είναι διαφορετική η προσέγγιση από αυτήν που έχει δώσει η Κομισιόν στην ετήσια έκθεση της Όλαφ. Είναι έκθεση δημοσιευμένη με στοιχεία δημοσιευμένα. Ε, πρέπει να πω ότι εμείς από την Κομισιόν έχουμε φτάσει σε πολύ πιο συνολικά συμπεράσματα βασιζόμενοι σε αυτά τα ποσοστά. Ε, γιατί εδώ ε, τεκμέρεται ότι το ποσοστό παρατυπιών είναι ίδιο σε όλες τις χώρες μέλη, πράγμα που ε, δεν ισχύει και επίσης δεν λαμβάνεται υπόψη το ειδικό οικονομικό ή άλλο περιβάλλον αναπερίπτωση για τις παρατυπίες. Θεωρούμε ότι επίσης ε, είναι μια υπερβολική προσέγγιση, προσέγγιση τύπου άσπρο-μαύρο, το να πει κανεί ότι το υψηλό ε, ποσοστό ανείχνευσης ε, παρατυπιών ταυτίζεται με ένα υψηλό επίπεδο ανάκτησης πόρων. Υπάρχουν, είναι πάρα πολλές οι χώρες οι οποίες παίρνουν μέτρα ε, και επομένως είναι λάθος να θεωρείται ένα χαμηλό ε, ποσοστό ανείχνευσης παρατυπιών σαν ε, μη ικανό σύστημα ή κακή επίδοση ας πούμε για τη Ρουμανία και χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες Ε, να πω ότι ας πούμε μια τόσο μικρή χώρα όσον αφορά τη συνεισφορά ε, πληρώνει παρόλα αυτά 2% των, ε, του ΑΕΠ σε ίδιους πόρους και επομένως αυτό μπορεί να θεωρηθεί ένα υψηλό ποσοστό ε, στατηγικά. Επίσης δεν θεωρούμε, δεν θεωρούμε σωστό το γεγονός ότι στην ε, μελέτη αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη ε, το η μακροπρόθεσμη δυνατότητα ανάκτησης πόρων. Και επίσης να σας πω ότι σε περίπτωση παρατυπιών το ποσοστό ανάκτησης εν τέλει φτάνει στο 20,4-20,5% ε, ε, και μάλιστα ε, την ίδια τη χρονιά ανείχνευση της παρατηρίας. Εάν δει κανείς ευρύτερη χρονική περίοδο 2006 ε, προκειμένου μέχρι 2011 ο βαθμός ανάκτησης ε, το ποσοστό ανάκτησης ε, των παρατυπιών φτάνει στο 70%. Η μελέτη δείχνει ότι το ποσοστό ανάκτησης για αυτές τις περιπτώσεις είναι 41%. Από τη δικιά μας πλευρά μακροπρόθεσμα αυτό το ποσοστό φτάνει στο 56%. Επομένως έχουμε μια αρκετά μεγάλη διαφορά με το ποσοστό το οποίο ε, αναγράφεται στην ε, μελέτη. Εδώ θα ήθελα επίσης ε, να παραθέσω την ανάλυση που είχαμε κάνει το 2009 και την αντίστοιχη ανάλυση της Όλαφ όσον αφορά το ιστορικό της ανάκτησης των παραδοσιακών πόρων. Αυτή η ανάλυση κατέδειξε ότι περίπου 80% των περιπτώσεων λύονται και επομένως τα ποσά ανακτώνται. Με αυτή την έννοια λοιπόν πιστεύω ότι η εικόνα που ε, μας έδειξε η Όλαφ όσον αφορά την ανάκτηση είναι σωστή. Επίσης ε, η προσέγγιση εδώ δεν ε, λαμβάνει υπόψη τις διαφορές προσέγγισης που έχουν τα κράτη-μέλη. Η κάθε χώρα έχει μια διαφορετική προσέγγιση, διαφορετική παράδοση αν θέλετε ανάκτησης των ιδίων πόρων και δεν σημαίνει ότι ένα μικρό λάθος ας πούμε στη δήλωση ε, ε, σημαίνει ταυτόχρονα ότι ανοίγουμε την πόρτα στους λαθρέμπορους. Αυτό που μας απασχολεί περισσότερο με την ε, προσέγγιση που παίρνει αυτή η μελέτη είναι αυτές ε, οι, αυτοί οι θεωρητικές δίκτες επίδοσης που έχουν καθοριστεί εν αγνία των ε, ε, στοιχείων ε, που πραγματικά ισχύουν σε κάθε χώρα. και με τον τρόπο αυτό ε, φτάνει σε ποσοστά ε, επίδοσης των κρατών μελών που δεν είναι σωστά και που βεβαίως ε, αντικρούονται από αξιόπιστες άλλες στατιστικές. Επίσης αυτό το ποσό των τριών δις δεν πείθομαι για το ποσό αυτό γιατί δεν βλέπω να υπάρχουν τα χειροπιαστά αποδεικτικά στοιχεία. Τέλος, ε, η ίδια η ομάδα των μελετητών φαίνεται ότι συμμερίζεται και τις δικές μας απόψεις γιατί επανειλημμένα λένε δεν γνωρίζουμε, δεν είμαστε σίγουροι. Και ε, όπως είπαν και οι ίδιοι στην ε, παρουσίαση που μόλις έκαναν, πρόκειται για, μια, για ένα θεωρητικό σχήμα και ακριβώς αυτή είναι και μια κριτική που ε, μπορώ να ασκήσω εγώ στο σύνολο της μελέτης αυτής. Τι κάνει η Κομισιόν για να βελτιώσει τις επιδόσεις των κρατών μελών. Πρώτα απ' όλα βεβαίως εστιάζουμε την προσοχή μας όχι στο 2% μονάχα, αλλά στο συνολικό ποσό. Ε, των παραδοσιακών ιδιών πόρων. Εμείς αποπτεύουμε ε, το σύνολο των παραδοσιακών ιδιών πόρων και θέλουμε να διασφαλιστεί η παράδοση του συνόλου των χρημάτων αυτών σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, και προβλέπουμε βεβαίως και μια ευρία γκάμα δράσεων. Τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να στείλουν όλα τα το σύνολο των ε, ποσών ε, που ε, προβλέπονται προς ανάκτηση και να δικαιολογούν με εκθέσεις τα ποσά αυτά, εκθέσεις τις οποίες μελετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μεταξύ του 6 και του 9 μελετήσαμε πάρα πολλές τέτοιες ε, ε, εκθέσεις ε, τις οποίες είχαμε λάβει από τα κράτη-μέλη και το 1 τέταρτο αυτών των 1.400 εκθέσεων αφορούσαν 1,5 δις ε, και βεβαίως ε, για αυτές, ε, για αυτές τις περιπτώσεις τα κράτη-μέλη οφείλουν να καταβάλουν τα χρήματα και όλη αυτή η διαδικασία στενά παρακολουθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βεβαίως γίνονται και οι απαραίτητες επιτόπου επιθεωρήσεις. So... I think this is very, very to, to, to... αυτός λοιπόν είναι ο τρόπος, ε, ο συγκεκριμένος τρόπος ε, μέσα από τον οποίο μπορούμε με συγκεκριμένο τρόπο λέω να αντιμετωπίσουμε τέτοια ζητήματα αποφεύγοντας υπερβολικές θεωρητικές προσεγγίσεις. και έτσι μας δίνεται και η δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε πραγματικά τις ε, αδυναμίες των κρατών μελών και τις ελλείψεις όσον αφορά την επίδοση των κρατών μελών. Επιπροσθέτως, Όπως ανέφεραν και οι ερευνητές, έχουμε και εμείς το δικό μας ε, σύστημα, τη δικιά μας ε, υπηρεσία ε, επιθεωρήσεων που στενά συνεργάζεται με τις επιτόπου αρχές οι οποίες είναι υπεύθυνες για την ανάκτηση παραδοσιακών πόρων. Και οπουδήποτε και οποτεδήποτε έχουμε ε, ταυτοποιήσει παρατυπία ή διοικητικό σφάλμα, ε, θεωρούμε το κράτος μέλος υπεύθυνο για την απώλεια. και αρκεί κανείς να περιτρέξει την νομολογία για να καταλάβει ότι υπάρχει ήδη ένα σύστημα υποστήριξης ε, με συγκεκριμένες δράσεις και με τις ε, δράσεις αυτές αποφεύγουμε ε, και ε, μεγάλες απώλειες ε, και πρόκειται για δράσεις τις οποίες εφαρμόζουμε σε όλα τα κράτη-μέλη. Επίσης, μεγάλη προσπάθεια καταβάλλεται σε σχέση με τις επιθεωρήσεις οι οποίες έχουν ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια και δίνουν και αποτελούν ένα καλό εργαλείο αξιολόγησης και διασφάλισης των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τις συστάσεις που γίνονται, πρέπει να πω ότι ήδη εποπτεύουμε τα patterns ανάκτησης των πόρων και τα αποτελέσματα δημοσιεύονται σε αιτήσια βάση. Επίσης λαμβάνονται υπόψη και κάποια διαρθρωτικά σχήματα, ε, structural patterns και επίσης ε, ε, μοιραζόμαστε με τα κράτη-μέλη τα αποτελέσματα και τα αναλύουμε και από κοινού έτσι ώστε να βοηθήσουμε και τα κράτη-μέλη να πάρουν τις σωστές αποφάσεις όσον αφορά τα προβλήματα. Φυσικά θα λάβουμε υπόψη τα ευρήματα ε, θα λάβουμε υπόψη ε, τις συστάσεις ε, της μελέτης, θα τις μελετήσουμε προσεκτικά. Αλλά για συγκεκριμένες δράσεις follow-up θεωρούμε ότι δεν μπορούν να βασιστούν σε τέτοιου είδους θεωρητικές ε, στατιστικές ε, ε, μελέτες και τέτοιου είδους στατιστικές θεωρητικές θεωρήσεις. Η Επιτροπή έχει ένα σύστημα ελέγχου το οποίο διαρκώς βελτιώνει και το οποίο βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. υπάρχει μια σύσταση ας πούμε στη μελέτη ότι θα πρέπει το ποσοστό να συνδέεται με την επίδοση. Να πω ότι για την ώρα δεν υπάρχει νομική βάση που να δικαιολογεί κάτι τέτοιο και επομένως θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε και συγκεκριμένα αξιόπιστα συγκριτικά στοιχεία που να μας οδηγήσουν σε αυτό το συμπέρασμα. Πιστεύουμε από τη δικιά μας πλευρά ότι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπιστούν οι πιθανές απώλειες που έχουν προκληθεί από τα κράτη-μέλη είναι να πληρώσουν τα ίδια τα κράτη-μέλη για τις απώλειες που έχουν προκύψει. Αυτά ήθελα να σας πω και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα δώσω λόγο αμέσως τον κύριο Γκάιερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ομολογώ ότι δεν έχω εγγύψει ας πούμε σε βάθος στον προβληματισμό αυτό. Περιθωριακά ασχοληθήκαμε στη συζήτηση των εκθέσεων απαλλαγής πρότεινα στην Επιτροπή και χαίρομαι που το δέχθηκαν και οι σκιώδεις να μην ασχοληθούμε μονάχα με την πλευρά των δαπανών αλλά και με το ερώτημα από πού έρχονται τα χρήματα και λαμβάνει άραγε η Ευρωπαϊκή Ένωση όλους τους πόρους που τις ε, αναλογούν σύμφωνα με τη συνθήκη στις συζητήσεις στο Συμβούλιο μπαίνει και το ερώτημα συνεχώς ποιος πληρώνει πόσα. Τα ποσά για τα οποία συζητούμε απέχουν πολύ από αυτά για τα οποία μάλωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και βέβαια και πολύ μακριά από αυτά που χρειάζονται για να κλείσουμε τον προϋπολογισμό του 2012. Αλλά τέλος πάντων Σωστό είναι να δούμε και λίγο ποιος εκπληρεί τα καθήκοντά του και ποιος ικανοποιεί τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Έχω μία ερώτηση τώρα προς τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, αλλά και προς τους ειδικού. Αν κατάλαβα καλά, οι συνεισφορές των χωρών μελών που δεν αποτελούνται ή προέρχονται από τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους, ζάχαρη, δασμούς κτλ. πρέπει να καλυφθούν από το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Άρα η χώρα μέλος η οποία δεν καταφέρει να κάνει optimal performance, άρεστη επίδοση με τους δασμούς, θα πρέπει να καλύψει το ελίπον από το ΑΕΠ. Άρα πρέπει να είναι και προς το συμφέρον των χωρών μελών να καλύψουν όσο γίνεται μεγαλύτερο ποσοστό από τους δασμούς. Διότι αλλιώς πρέπει να τα καλύψουν από το ΑΕΠ και νομίζω ότι ούτως ή άλλως κρατά και 20% των ιδίων πόρων, των παραδοσιακών ιδίων πόρων η χώρα μέλος ως handling fees, ως τέλη χειρισμού. Θα, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να ικανοποιήσει αυτός του δημοσιογράφου, αλλά εν πάση περιπτώσει θέτω το ερώτημα. Δεύτερο, ποια είναι η αναλογία με τα δηλωμένα ποσά των δασμών που ωστόσο δεν έχουν εισπραχθεί από τις χώρες μέλη. Ποια είναι η σχέση λοιπόν αυτή με το συνολικό όγκο του εμπορίου. Δηλαδή, σκοπό να καταλήξω σε μια ερώτηση που έχει απασχολήσει ήδη την Επιτροπή μας και μάλιστα και σε μια αντιπροσωπεία στα λιμάνια του Ρότερνταμ και της Αμβέρσας. Λαμβάνουμε πράγματι από τις χώρες μέλη τους δασμούς στο ύψος που μπορούμε να τους λάβουμε. Νομίζω ότι αυτό δεν το έχει μελετήσει ούτε η ίδια η μελέτη. Διότι αν κατάλαβα καλά, το πεδίο εφαρμογή της μελέτης περιορίστηκε μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που έχουν, δηλαδή τα έσοδα εκείνα από δασμούς που έχουν δηλώσει οι χώρες μέλη. Δηλαδή δεν εγκύψατε στον προβληματισμό ή τέλο πάντων δεν έχετε συλλέξει στοιχεία σχετικά με το αν πέραν αυτών αν ενδεχομένως δεν δουλέψει καλά το τελωνίο, τι γίνεται. Και τέλος, προς τους ειδικού γράφετε συστάσεις και για την Κομισιόν και για τις χώρε μέλη. Ναι, αλλά πού θα τα συζητήσουν, πού θα συζητήσουν αυτές τις συστάσεις οι χώρε μέλη. Μήπω πρέπει να γράψετε συστάσεις προς το Συμβούλιο. Ως πολιτικός, εγώ προσωπικά αντιμετωπίζω πάντοτε το πρόβλημα ότι δεν μπορώ να αρπάξω πουθενά τι χώρε μέλη. Δεν μπορώ να τι τριμώξω πουθενά. Εκπλούν τα καθήκοντά του, πότε καλύτερα, πότε χειρότερα, συνήθω χειρότερα και το Συμβούλιο απέναντι στην Κομισιόν συστήνει την απαλλαγή, δεν κάνει όμως κρίση ομοτήμων, peer review μεταξύ τους, οι χώρες μέλη, δεν κάνουν για το αν κάνουν καλύτερα ή χειρότερα τη δουλειά τους. Βέβαια πρέπει να είναι διπλωματικές οι χώρες μέλη μεταξύ τους, τι να πω, ας το πω κοινικά ή ίσως και σαργαστικά, αλλά ίσως έχουμε και κάποια προβλήματα να πούμε σε κάποια χώρα μέρος κοίτα να δεις θα μπορούσε να κάνεις και κάτι καλύτερο. Αλλά δεν ξεφεύγουμε από το πρόβλημα, εάν οι χώρες μέλη ή οι ίδιες αντιμετωπίζουν οι μεν τις δε σαν να βρισκόμαστε στο χείλο του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου και άρα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά διπλωματικοί, τότε ίσως δεν έχουμε και περιθώριο να παίξουμε διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να επισημαίνει τι ευθύνε των χωρών μελών, οι χώρε μέλη δεν δέχονται τίποτα και το Συμβούλιο δεν υιοθετεί τη συζήτηση, αλλά πετάει τον μπαλάκι παραπέρα στην Κομισιόν. Η Κομισιόν βεβαίω ζητούμε να κάνει καλύτερη τη δουλειά, τη δουλειά της και βεβαίω οι αξιωματικοί τη Κομισιόν θέλουν, αλλά δεν έχουν τον απαραίτητο εταίρο που θα ήταν το Συμβούλιο. Ίσως μπορεί να τοποθετηθεί και πάλι ο εκπρόσωπος της Κομισιόν δεν είναι ανάγκη να μου πει κύριε Γκάιερ έχετε δίκιο γιατί η παρατήρηση που έκανα ήταν κάπως σαρκαστική αλλά αν κατανόησα καλά το πρόβλημα τότε θα ήμουν ευγνώμων πάντως να ακούσω μια άποψη. Ευχαριστώ, δεν έχω άλλα σχόλια και γι' αυτό προτείνω να δώσουμε το λόγο και πάλι στην Κομισιόν ώστε ο εκπρόσωπός της να απαντήσει στον κύριο Γκάιρ. Καλά λοιπόν. Αλλά πρώτα η κυρία Ντελάγκε και μετά η Κομισιόν να απαντήσει σε ένα δίλεπτο. Είδε ειδικοί να τοποθετηθούν μέσα σε ένα διάστημα τεσσάρων λεπτών. Και θα δώσω πάλι το λόγο στην κυρία Ντελάγκε. Ευχαριστώ πριν πάει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και βέβαια αυτό είναι πρότυπο ή μοντέλο, δεν ξέρω, και πάντα υπάρχουν αποχρόντες λόγοι, γιατί η πραγματικότητα είναι πολύ περίπλοκη από ένα μοντέλο. Αλλά τουλάχιστον έχουμε αυτό το μοντέλο. Εγώ είμαι πέντε χρόνια μέλος εδώ και αυτό που ακούω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να το κοιτάξουμε ad hoc, ένα περίπτωση. Όταν έχει ένα μοντέλο όμω μπορεί να εντοπίσει διαχρονικά κάποιου δείκτε, κάποιε τάσει Γι' αυτό το θεωρώ ενδιαφέρον. Και έχω δύο συγκεκριμένε ερωτήσει να κάνω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι οποίε μπορεί να απαντήσει με ένα ναι ή με ένα όχι. Υπάρχουν διαφορέ μεταξύ των κρατών μελών στι επιδόσει του. όταν πρόκειται για την ανάκτηση ε, πόρων και ποσών από τους ε, παραδοσιακούς ιδίους πόρους. Ναι, Ερώτηση δεύτερη. Είναι προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κινηθούμε όλοι ε, προς ε, τις άριστες επιδόσεις όσο γίνεται να τις προσεγγίσουμε. Ναι, Δύο ερωτήσεις με πολύ απλή απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ιδιαίτερα όταν βλέπω ποσά που θεωρητικά θα πρέπει να πηγαίνουν τα ποσά αυτά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά παραμένουν προς το παρόν σε επίπεδο κρατών μελών. 30% του λογαριασμού Β ε, είναι σε ένα κράτος μέλος. Ρωτώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχουν διαφορές στις επιδόσεις των κρατών μελών εδώ, νέου και είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κινηθούμε όλοι μαζί προς μια βέλτιστη πρακτική προς τις άριστες επιδόσεις, αντί απλώς μυρολατρικά να δεχόμαστε ότι υπάρχουν διαφορές. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος. Θα δώσω το λόγο τώρα στον ε, πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Δύο λεπτά και μετά η δική μας ε, ε, για άλλα τέσσερα λεπτά, όπως είπαμε, για να κλείσει αυτό το θέμα. Τελευταία θα ξαναπάρει το λόγο η συγγήτρια για να συνοψίσει. Δεν θέλω, λέει η κυρία Ντελάνγκιο. Sorry, micro, please. First for the question. Πρώτα, για την ερώτηση για τους πόρους που δεν εισπράττονται από τις χώρες μέλη. λόγω μη επιμελούς δράσης. Είναι αληθές ότι λόγω του ισορροπημένου συστήματος για τον κοινοτικό προϋπολογισμό όσα ποσά δεν εισπραχθούν από τους ε, ε, δασμούς τους, δηλαδή παραδοσιακούς σπόρους δηλαδή, πρέπει να καλυφθούν από το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. οι δεμοί θα πρέπει να μοιραστούν το βάρος και άλλες φορές. Και γι' αυτό έχουμε την προσέγγιση της οικονομικής ευθύνης. στην δραστηριότητα ελέγχου μας απέναντι στις χώρες μέλη. Αυτή τη στιγμή δηλαδή εντοπίσουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, ένα συγκεκριμένο λάθος, είτε πρόκειται για διαθροτικό είτε πρόκειται για ατομικό. Ζητούμε από τη χώρα μέλος να καταβάλει το σχετικό ποσό. Δεν συμφωνούν πάντα οι χώρε μέλη με την προσέγγιση αυτή και έχουμε κατ' επανάληψη προσφυγέ στα δικαστήρια. Το δικαστήριο όμω επικύρωσε την προσέγγιση μα. Και αυτό είναι ο δρόμο που οφείλουμε να ακολουθήσουμε. Μέσα όμως στο παρόν πλαίσιο δεν μπορούμε να προσφύγουμε κατά των χωρών μελών για να απαιτήσουμε καταβολή ποσών στη βάση στατιστικών. Έχουμε τα ετήσια προγράμματα ελέγχων και σε αυτά βασιζόμαστε. Αλλιώ, όπω είπα, άλλε χώρε μέλη θα χρειαστεί να συμβάλλουν για να αντιμετωπιστούν τα κενά, να πληρωθούν τα κενά. Διαφορέ στην επίδοση. Ναι, βεβαίω υπάρχουν. Οι χώρε μέλη είναι διαφορετικέ, οι εθνικέ διαδικασίε είναι διαφορετικέ, οι διοικήσει είναι διαφορετικέ. Δεν θα βρείτε δύο χώρε μέλη που να έχουν ακριβώ την ίδια επίδοση. Πάντα υπάρχουν διαφορέ. Δεν συζητώ τώρα για το εάν από τις διαφορές αυτές προκύπτει η διαφορά των ποσών που διαλαμβάνει η μελέτη. Εάν διαπιστώσουμε πάντως διαφορές που δείχνει μη επιμελή δράση των χωρών μελών, τότε απαιτούμε την εισπράξη των ποσών. Έτσι αντιμετωπίζουμε τα θέματα αυτά. Οι αναλυτικές μελέτες έχουν ενδιαφέρον, αλλά το μόνο που μπορούν να κάνουν να προσφέρουν ιδέες για στόχευση των δράσεων ελέγχων. Δεν μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για συγκεκριμένες δράσεις. Για συγκεκριμένες δράσεις χρειαζόμαστε και συγκεκριμένα πορίσματα ελέγχων. Εξάλλου, ναι. Θα ήταν πολύ χρήσιμο αν όλες οι χώρες μέλη μπορούσαν να αποδίδουν στο επίπεδο του best performer, της χώρας που αποδίδει καλύτερα. Εμείς έχουμε προσφέρει, έχουμε διαβάσει τις χώρες μέλη κείμενα με τις αρχές που εφαρμόζουν οι χώρες που έχουν τη μέγιστη ε, απόδοση και αυτό ζητούμε να ακολουθήσουν. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Εσείς παρακαλώ. I'd like to start and then I'll pass the... Επιτρέψτε μου να αρχίσω και μετά να συνεχίσω ο συναδελφός μου. Χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει καλά τις στατιστικές που δημοσιεύει και που προσπαθεί να τις χρησιμοποιήσει συστηματικά με την βοήθειά μας. Και συγχαίρω την Επιτροπή που το πράττει αυτό. Είμαι λίγο απογοητευμένος για το γεγονός ότι δεν κατέστησαν ωστόσο ικανοί να καταλήξουν στις, στα συστημικά συμπεράσματα στα οποία καταλήγουμε εμείς. Αφού υπάρχει το 2% που διαφεύγει. Και είναι πάντως ένας αριθμός σχετικά μεγάλος, δηλαδή είναι περίπου 3 δισεκατομμύρια. Και 3 δισεκατομμύρια, όπως και να το δει κανείς, είναι πολλά λεφτά. Δεύτερο, υπάρχουν συνθήκες υπό τις οποίες συζητούν χωρίς μέλη και κομισιόν για τα θέματα αυτά. Στην Επιτροπή Ιδιών Πόρων, για παράδειγμα. Όμως δεν είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς τι διαμείβεται σε αυτές τις συζητήσεις. Η δική μου εμπειρία μου δείχνει ότι είναι μάλλον διπλωματικές υποθέσεις αυτές και όχι η αντιπαράθεση που θα ανέμενε κανείς να είναι, ιδίω όταν υπάρχουν σημαντικές, προφανώς σημαντικές διαφορές απόδοση μεταξύ των χωρών Το θέμα είναι στην ουσία η μεταφορά των πληρωμών από τους οικονομικούς φορείς η μεταφορά από, την οικονομία, από, αυτά που, χρωστά, θα χρωστούσαν κανονικά οικονομικό περίπτωση τα καλύπτουν τελικά οι φορολογούμενοι. Και εγώ νομίζω ότι αυτό είναι μια έμεση επιδότηση. Επιτρέψτε μου να παραδώσω το μικρόφωνο στον Ντέιβιτς που θα επισέλθει σε πιο ειδικά θέματα. Αλλά επισημαίνω την προσοχή σας σε μία από τις συστάσεις που εξακολουθεί να ισχύει ότι μπορεί να θεωρήσει κανείς το 20% των χωρών μελών που, που, που κρατούν μάλλον οι χώρες μέλη ως τέλη χειρισμού ότι αυτό θα μπορούσε το ποσό αυτό να καταστεί εύκαμπτο με την έννοια ότι θα μειώνεται εάν δεν είναι ικανοποιητική η επίδοση της χώρας. Και νομίζω ότι αυτό είναι ε, ένα μονοπάτι ενδιαφέρον να το διαβεί κανείς. Ευχαριστώ. Πρόσθετες παρατηρήσεις για τα δεδομένα που χρησιμοποίησαμε. Όντως βασίστηκαν σε, βασίστηκε σε, αυτή, σε αυτά τα ε, δεδομένα ένα θεωρητικό εγχείρημα. Είναι όμως δημόσια δεδομένα ή δεδομένα τα οποία ζητήσαμε και λάβαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το μόνο που κάναμε ήταν να συνδυάσουμε τα δεδομένα αυτά ανοιχτή πηγή με αυτά τα ενδιαφέροντα σχήματα τα οποία προκύπτουν. Και όχι μόνο στο έτος αναφοράς, αλλά εμεί προχωρήσαμε σε μια μελέτη έξι ετών. Και από αυτά τα ενδιαφέροντα σχήματα που είπα πριν, τα patterns αυτά, δεν θα μπω λοιπόν πολύ στα τεχνικά θέματα, γιατί όπου υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα και ενδέχεται να επηρεάσουν τα αποτελέσματά μας, θα πήραμε υπόψη. Άκουσα μια παρατήρηση για ιστορικό ρεκόρ απόδοσης. Μας ενδιαφέρει πολύ γιατί θα μας έδειχνε την βέλτιστη εικόνα της απόδοσης μιας χώρας στην ανάκτηση. Αλλά από τα έξι χρόνια που κοιτάξαμε, πέντε από τις σχετικές εκθέσεις της Όλαφ περιλαμβάνουν τέτοιο ιστορικό ε, επίπεδο. Η μία όμω όχι. Αλλιώ θα θέλαμε να τα χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά. Πάντως, φτάσαμε μέχρι να πούμε, καλά, θα πάρουμε το recovery rate ενό έτου, αλλά φανταστείτε να είναι α πούμε 70% ή 80% όπω είπαν ορισμένοι. Ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα. Εν τέλει θα ήταν 600 εκατομμύρια. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ του ποσού που έχει ήδη καλυφθεί, το 43% και το 80%. Θα μείωνε λοιπόν τα συμπεράσματά μας κατά λίγο πάνω από μισό δισεκατομμύριο. Δεν θα άλλαζε δηλαδή πολύ σοβαρά τα συμπεράσματά μας. Τρίτο, πιο σημαντικό ίσως. Είπαμε ότι αυτό που κάνει η Κομισιόν είναι πολύ θετικό. Διότι όταν διαπίστωσαν ζημία του κοινοτικού προϋπολογισμού, επεβάλλουν κύρωση σε αυτούς που έφτυγαν με τις αποφάσεις. Αυτό που κάναμε εμεί ωστόσο στο δικό μας εγχείρημα ήταν να χρησιμοποιήσουμε στατηγικά δεδομένα για να δείξουμε τι ενδεχομένως δεν έχουν κάνει οι χωρισμένοι. Και δεν μπορεί κανείς να βρει τέτοια ζημία στον προϋπολογισμό ε, στοχεύοντας μόνο σε οικονομικούς ελέγχους, επιθεωρήσεις κλπ. Αν πάρετε λοιπόν τα δεδομένα σε μεγαλύτερο, σε ευρύτερο πλαίσιο, και αυτό κάναμε, μπορείτε να στοχεύσετε στο τι δεν έπραξαν οι χώρε μέλη, ενώ θα έπρεπε να είχαν πράξει. Και εκεί προσπαθήσαμε να καταλήξουμε σε κάποια εκτίμηση που όντω είναι θεωρητική, αλλά είμαστε βέβαιοι ότι αν εξετάσετε το τι θα έπρεπε να είχαν κάνει οι χώρε μέλη και προσπαθήσετε να ε, το υπολογίσετε θα βρείτε κάτι διαφορετικό. Και απαντώ τώρα στην ερώτηση της κυρίας Λάνια είναι ενδιαφέρον ως μοντέλο να αξιολογήσουμε άλλες εκτιμήσεις στο δημοσιονομικό πεδίο. Προσπαθήσαμε στην αρχή, είχαμε μια προκατακτική μελέτη που έδειχνε ότι υπήρχαν διαφορές. Όταν αρχίσαμε το εγχείρημα, διαπιστώσαμε διαφορές παντού και μάλιστα ουσιαστικές και διαστοτικές όταν διαπιστώσαμε ποιοι ήταν οι λόγοι για τις διαφορές αυτές, δηλαδή οι διαφορές μεταξύ των χωρών μελών στην ανάκτηση σε περιπτώσεις ατασταλιών, ενώ όπου δηλαδή οι χώρες μέλη πρέπει να κάνουν το ίδιο πράγμα, διαπιστώσαμε ότι αυτό μπορεί να προσαρμοστεί και σε άλλους τομείς του προϋπολογισμού. Το κάναμε αυτό για τον τομέα των τελωνίων, που για τα έξι χρόνια ανέρχεται σε 127 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή περίπου 22 ευρώ τον χρόνο, 22 συγγνώμη, δισεκατομμύρια τον χρόνο. Πώς θα απέδει το μοντέλο αυτό, αν αυτό ε, εφαρμοζόταν και στο indirect expenditure στις έμεσες δαπάνες. Εκεί είδαμε ότι τα ποσά θα ήταν πενταπλάσια. Μιλάμε για 100 δισεκατομμύρια, αλλά τα φαινόμενα που φαίνεται να λαμβάνουν χώρα στον τομέα των εσόδων είναι παρόμοια. Βέβαια, τεχνικά δεν μπορούμε να απαντήσουμε στην ερώτηση, αλλά ίσως αυτά που βρήκαμε στα έσοδα, ίσως να ανέρχονται στο πενταπλάσιο των όσων βρήκαμε στον τομέα των δαπανών, στην πλευρά των δαπανών. Γιατί ο χειρισμός των έμεσων δαπανών γίνεται από τις αρχές των χωρών μελών. Και αν εξετάσετε τις ατα, που μπορούν να βρεθούν και στις ίδιες εκθέσεις της όλα, θα βρείτε τους ίδιους μηχανισμούς. Πιστεύουμε λοιπόν σίγουρα ότι αυτό μπορεί να εξυπηρετήσει, μπορεί να ωφελήσει και στον δημοσιονομικό τομέα. Και μια τελική παρατήρηση για το πώς μπορεί κανείς να το δει, να το εξετάσει έγινε μια παρατήρηση για την κατάσταση στο Βέλγιο και στην Ολλανδία. Διότι ε, ταξιδεύσατε, πήγατε στη Ρότερνταμ και στην Αμβέρσα. Θα είδατε ότι η κατάσταση αυτή είναι παρόμοια. Δύο μεγάλα λιμάνια μικρών χωρών με παρόμοια οικονομικά συστήματα λίγο πολύ. Και κοιτάξτε τις διαφάνειες μας στο detection stage θα δείτε τεράστιες διαφορές στα αποτελέσματα που έχουμε αποκάλυψης, detection και για τις βελικές και για τις ολλανδικές αρχές. Αυτό μπορεί να ισχύσει για όλες τις φάσεις και για όλα τα θέματα. Με αυτό θα ήθελα να ολοκληρώσω εδώ την παρουσίασή μας, γιατί ελπίζω ότι το παράδειγμα αυτό πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Αγαπητοί συνάδελφοι, ολοκληρώνεται εδώ αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης και παίρνουμε στο επόμενο. Ταμείο ενίσχυσης των απόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι γνωμοδότηση αυτή, γιατί δεν είμαστε αρμόδιοι επί της ουσίας. Συντάκτης είναι ο κύριος Σεόδωρος Κυλακάκης, ο οποίος μας ε, διαβίβασε ότι έχει άλλες ανηλμένες υποχρεώσεις και ακολύεται σήμερα. Επειδή δεν έχουμε και χρόνο, πρέπει να σας πω δε ότι υπάρχει μόνο στα αγγλικά η γνωμοδότηση και θέλω να ρωτήσω τους συναδέλφους αν υπάρχει κανείς που έχει να κάνει ερωτήσεις ή παρατηρήσεις για τη γνωμοδότηση αυτή που υπάρχει μόνο στα αγγλικά. Δεν ζητεί κανείς να έρθει στο λόγο. Και θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών έχει οριστεί για την 22η Μαρτίου 2013 και ώρα 12η μεσημβρινή. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, Συνεχίζουμε και παίρνουμε στο επόμενο σημείο στη μέση διάταξη που είναι... Ε, Μα ζητώ συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος. Έχουμε ένα μικρό τεχνικό διάλειμμα, μια μικρή διακοπή. Okay. Ah, uh, oh, sorry. Please uh, stay there. Szóval, tisztelt képviselőtársaim! Λοιπόν, έλεγα αγαπητοί συνάδελφοι ότι ε, θα περάσουμε τώρα στο σημείο υπαριθμών 58 και θα έχουμε συζήτηση με τον κύριο Χέρμπερτ Μπέρς. Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Όλαφ. Κύριος Μπέρς είναι πρώην συνάδελφος, πρώην μέλος της Επιτροπής μας. Σας καλωσορίζω θερμά στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. και μάλιστα έχετε διατελέσει και πρόεδρος της Επιτροπής Ελεγχού Προϋπολογισμού. Σας παρακαλέσαμε να έρθετε εδώ στο Προεδρείο, αλλά μας είπατε ότι δεν επιθυμείτε να μιλήσετε από εδώ. Σας δίνω μέσα στο λόγο για να μας κάνετε μια παρουσίαση για το θέμα αυτό. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λειτουργεί το μικρόφωνο, ε, μάλιστα. Ε, ε, σας ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Με μεγάλη χαρά ήρθαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να σας μιλήσουμε για την αναθεώρηση, τροποποίηση του κανονισμού για την Όλαφ και να σας δώσουμε τις δικές μας απόψεις. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση διότι γνωρίζουμε βεβαίως ότι εδώ και χρόνια είναι αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Έχουμε καθυστερήσει λίγο σε σχέση με τον παλαιό κανονισμό που είχε προβλέψει μια τριετή ε, φάση. Πάντως υπάρχει και ένας άλλος λόγος που χαιρόμαστε που ήρθαμε εδώ στο Κοινοβούλιο το οποίο βεβαίω σεβόμαστε, δεν είναι μόνο λόγο σεβασμού, αλλά θέλουμε να ενημερώσουμε και το Κοινοβούλιο για το πώς βλέπουμε εμείς τα πράγματα. Είμαστε νεοσύστατη επιτροπή, ένα χρόνο είναι η ζωή της επιτροπής μας, να δούμε τι συμπεράσματα έχουμε βγάλει από τις παρατηρήσεις όσο και τις ε, έρευνες σε διάφορες περιπτώσεις και πολλές υποθέσεις για να δούμε πώς θα πρέπει να διαμορφωθεί ο νέος κανονισμός ή το σχέδιο που διαπραγματεύονται τα θεσμικά όργανα μεταξύ τους. Είναι και το λεγόμενο ISIP, που σημαίνει ε, εντολές προς το προσωπικό ε, και διαδικαστικές ρυθμίσεις. Ήταν το προηγούμενο εγχειρίδιο το οποίο αντικαθίσταται από τις νέες διατάξεις και να επισημάνουμε κάποιες ε, αδυναμίες και κάποια ισχυρά δυνατά σημεία. Λοιπόν, γνωρίζετε ότι μας υποχρεώνει η συνθήκη ε, σε αιτήσια βάση να καταθέτουμε έκθεση. Αποφασίσαμε λοιπόν ένα τμήμα της ετήσιας έκθεσης να το αφιερώσουμε σε αυτόν ακριβώς τον τομέα. Και γι' αυτό συντάξαμε ένα έγγραφο εργασίας. Θα ήθελα να σας ενημερώσω έτσι, με κάποια αποσπάσματα. Έχουμε ενημερώσει και τον αρμόδιο επίτροπο σχετικά ότι αυτές είναι οι προθέσεις μας. Αν με ρωτούσε τώρα κάποιος πώς βλέπω τον κανονισμό και τι φρονώ για τον κανονισμό που θα πρέπει να αποφασιστεί. Πρέπει να σας πω συντάκτης του εγγράφου εργασίας ότι βλέποντας και κάνοντας που ξέρω ότι εσείς στο Κοινοβούλιο ε, έχετε την κυριαρχία να το διαπραγματευτείτε. Να σας πω γιατί το λέω αυτό. Στάση αναμονής. Εμείς καταβάλαμε την προσπάθεια να στείλουμε τις εκθέσεις μας, μία από τις εκθέσεις μας και στο Κοινοβούλιο. Και νομίζω ότι χρειάζεται μελέτη αυτή η έκθεση πριν αποφασιστούν νέα μέτρα για την τροποποίηση και τη μεταρρύθμιση της υπηρεσίας τα πολέμες της απάτης, όλα και εδώ πρόκειται για ένα χρονικό ορίζοντα αρκετά ε, λογικό και θα άξιζε τον κόπο η ετήσια έκθεση που ελπίζουμε να εγκρίνουμε τον Απρίλιο συμπεριλαμβανομένου του παρόντος εγγράφου εργασίας να ε, αποτελέσει αντικείμενο ανάλυσης της μεταρρύθμισης και να ληφθεί υπόψη πριν ε, ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση. Τουλάχιστον να έχετε λάβει γνώση, να έχετε μελετήσει το έγγραφο αυτό. Θα προσπαθήσω τώρα με τα καλύτερα αγγλικά μου να σας διασκεδάσω, διότι τα λέμε στα αγγλικά αυτά, ε, τα γράφουμε στα κείμενά μας. Να σας πω τι μας απασχόλησε στο έγγραφο εργασίας. Και ε, ζητώ και πάλι συγγνώμη, δεν σας έχουμε διαβάσει ακόμα το έγγραφο αυτό γιατί δεν έχει αποφασιστεί ακόμα επίσημα από το σύνολο της Επιτροπής μας. Λοιπόν, στα αγγλικά τώρα, τι κοιτάξαμε. Τα μέτρα ε, ερεύνης που έχει δικαίωμα να λάβει η Όλαφ, πρώτον. Δεύτερον, το σεβασμό των ε, δικαιοδοτικών ε, αρμοδιοτήτων, της έρευνε της ΟΛΑΦ με σεβασμό το δικαίου των κρατών μελών, ε, η διάκριση των ερευνών εσωτερικές εξωτερικές, άμεση συμμετοχή του Γενικού Διευθυντού της Όλαφ σε ε, ερευνητικές δραστηριότητες, ε, προτεραιότητες πολιτικής και η έννοια της επαρκούς υποψίας αναθεώρηση των δράσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Όλαφ, η διαφορά μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών ερευνών και ο ρόλος της Εποπτικής Επιτροπής μας ε, στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της σωστής διεξαγωγής των ερευνών της Όλαφ. Λοιπόν, δεν θα τα παραθέσω όλα στα αγγλικά, αλλά ενδεχομένως δύο-τρία σημεία ακόμα, αν μου επιτρέπετε. διοικητικές έρευνες και ερευνητικά μέτρα που ε, επιτρέπεται να λαμβάνει όλα. Επαναλαμβάνω και πάλι, αυτό είναι το αποτέλεσμα πολλών ε, ερευνών που κάναμε στην Επιτροπή μας ε, το τελευταίο έτος. Στο άρθρο 2 του κειμένου του κανονισμού 1073 του 99 λέγει ότι ε, διοικητικές έρευνες σημαίνουν επιθεώρηση, έλεγχο ή άλλα μέτρα που κάνει η Όλαφ ε, βάσει των άρθρων 3 και 4. Τι λέγουν τα άρθρα 3 και 4. Έχουν ένα εξαντλητικό ε, κατάλογο μέτρων ερευνητικών και αντιστοιχεί το κείμενο με το άρθρο 2 του κανονισμού που ισχύει σήμερα το άρθρο 11.5 των IC, που όπως κυκλοφόρησε από το Γενικό Διευθυντή της Όλαφ, δείχνει ποια είναι τα μέσα ε, που έχει στη διάθεσή της Όλαφ για να συλλέγει ε, στοιχεία. Αυτά περιλαμβάνονται στα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού. Ωστόσο, αυτή η διάταξη ε, δεν θεωρεί τον κατάλογο αυτό εξαντλητικό, διότι αναφέρεται ότι είναι μεταξύ άλλων τα μέτρα αυτά, είναι τεράλια.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 Από την ελεγκτική λοιπόν δραστηριότητα που έχει δική μας επιτροπή μπορούμε να πούμε ότι η Όλαφ έχει αναλάβει ερευνητικά μέτρα που υπερβαίνουν το πλαίσιο των άρθρων 3 και 4 του ισχύοντος κανονισμούς και υπερβαίνουν και το μελλοντικό κείμενο της ε, αναθεώρησης. Μεταξύ άλλων να προετοιμάζει και να βοηθάει στην ε, μαγνητοφώνηση μιας ιδιωτικής τηλεφωνικής συνδιάλεξη; Μα δεν απορρέει από το κείμενο του κανονισμού, ούτε υπάρχει ειδική νομική ανάλυση που να έχει κάνει όλα Όλαφ πριν εκτελέσει αυτό το μέτρο. Και τα δύο αυτά είναι ερευνητικά μέτρα που μπορούν να θεωρηθούν επέμβαση δημόσιας αρχής ε, και ε, ε, στην ιδιωτική ζωή και στην αλληλογραφία που κανονικά αυτά διέπονται από την νομοθεσία άρθρων 7 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιστοιχεί στα όσα εγγυάται και το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΕΣΔΑ. Παρά την αιτιολογική σκέψη του 18 της μεταρρύθμισης που λέγει ότι οι κατευθυντήρες γραμμές ε, του Γενικού Διευθυντή της Όλαφ δεν θα πρέπει να δημιουργήσουν ή να ε, αλλοιώσουν οποιοδήποτε δικαίωμα απορρέει από το παράγοντα κανονισμό. Ενδεχομένως υπάρχει μεγάλος κίνδυνος όμως ε, και η Επιτροπή μας η Εποπτική θεωρεί ότι θα ήταν σημαντικό να διευκρινιστεί εκτενώς η φύση των ερευνών στο κείμενο της τροποποίησης του κανονισμού. Θα μπορούσα να σας αναφέρω και ένα δεύτερο σημείο αναφορικά με αυτό. Εν πάση περιπτώσει θα σας διαβεβάσουμε το κείμενο όπως σας είπα σε απότερο στάδιο. Όταν εγκριθεί η άμεση συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή της Όλαφ στις δραστηριότητες ερευνητικές της Όλαφ υπό τον παρόντα κανονισμό Γενικός Διευθυντής ε, διεξάγει τις έρευνες και καταρχήν ε, στην τροποποίηση διατηρείται αυτό και η έρευνα θα πρέπει να γίνει υπό τη δική του διεύθυνση από τους υπαλλήλους που έχουν οριστεί από τον ίδιο. Και αυτά τονίζονται στην αιτιολογική σκέψη 19. Το προσωπικό της Όλαφ καλείται να ασκεί τις έρευνες βάσει των κατευθυντηρίων γραμμών για τις διαδικασίες και βάσει μεμονωμένων και ατομικών εντολών που, και υποδείξεων που δίνει ο Γενικός Διευθυντής ε, σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Και πάλι βάσει τη εμπειρία η Επιτροπή μας ανησυχεί για την άμεση συμμετοχή του Γενικού Διευθυντού σε δραστηριότητε, όπως είναι συνεντεύξει μαρτύρων και προσώπων ε, ενεχομένων και επιτοπίων ελέγχων τίθεται ένα ζήτημα εδώ. Ο ίδιος ο Γενικός Διευθυντής Αυτοπροσώπος συμμετέχει στις έρευνες. Αυτό είναι σημαντικό ερώτημα. Και αυτό θα ε, μπορεί να επηρεάσει την αρχή της ε, αμεροληψίας σε εσωτερικές έρευνες. Ιδιαίτερα ε, στο άρθρο 90α του υπηρεσιακού του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης ορίζεται ότι οποιοδήποτε ελεγχόμενος μπορεί να υποβάλει στον Γενικό Διευθυντή της Όλαφ ε, καταγγελία ή παράπονο για ένα θέμα που τον θίγει ε, από τις έρευνες που διεξάγει Όλαφ. Η Εποπτική Επιτροπή λοιπόν θα ήθελε να τονίσει ότι η νομολογία έχει δώσει ένα, ορισμό, ένα γενικό ορισμό στο θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων και θεωρεί ότι ο Γενικός Διευθυντής καλό θα ήταν να μην μπαίνει στον κίνδυνο να ε, φέρεται σε μια ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων που θα διακύβευε και την αναθεώρηση των δράσεων της Όλαφ. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια σαφής διατύπωση στον τροποποιημένο κανονισμό σχετικά. Γνωρίζω ότι θα πρέπει να γίνει και συζήτηση κύριε Πρόεδρε και δεν θέλω να ε, μακρηγορήσω και να συνεχίσω να σας εξηγώ ε, τη σκέψη μας. Σας είπα τον Απρίλιο θα εγκριθεί το κείμενο στο σύνολό του. Απλώς ε, υπάρχει ένας ολόκληρος κατάλογος σοβαρών όμως ανησυχιών μας σχετικά με τα σημεία που ερευνήσαμε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Μπες. Ευχαριστώ για την ανάπτυξη των σκέψεών σας. Η κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ. Επισημαίνω το εξής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από όθηση της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού ζήτησε έκθεση της Εποπτικής Επιτροπής για την υπόθεση Ντάλι. Η έκθεση αυτή υπάρχει από την 21η Πρώτου. Τηρείται απόρριτη. Αυτοί που την τηρούν απόρριτη αποδέχονται και καλύπτουν παραβίαση του δικαίου. Προφανώς, είναι προφανής η παραβίαση του δικαίου όταν ακούω ότι οι ιδιωτικές τηλεφωνικές συνομιλίες παρακολουθούνται και μάλιστα ακούγονται και συμβουλές για το πώς μπορεί να γίνει καλύτερα. Ποια είναι η έννοια της έρευνας να συλλεχθούν οι υφιστάμενες αποδείξεις. Η έννοια της έρευνας είναι η συλλογή ενοχοποιητικού ή αθωτικού υλικού. Όταν ακούω ότι γίνονται τέτοια τηλεφωνήματα, δεν είναι δυνατόν παρά να κατασκευάζονται τέτοια ενοχοποιητικά στοιχεία. Τα έχετε δει αυτά κύριε Μπέσ στην εργασία που έχετε αναλάβει. Ότι κατασκευάζονται αποδείξεις. Θέλω να το μάθω αυτό. Δεύτερο, αυτή η παρακολούθηση και καταγραφή τηλεφωνημάτων. Πώς τα κρίνει η Εποπτική Επιτροπή σας. Εμείς ακούμε ότι πρόκειται για παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου και του δικαίου της προστασίας των δεδομένων. Ακούμε ότι έχει σχέση με θεσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φαίνεται ότι δρά απολύτως ανεξάρτητα από χώρο και χρόνο. Καλά τα έχω μάθει και καταλάβει αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ κύριος Γκάιερ. Η παρέμβασή μου θα είναι κάπως μακρά, διότι θέλω να εξηγήσω ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Εμείς διαπραγματευτήκαμε κανονισμό για την Όλαφ σε τριμερή διάλογο και με συμμετοχή όλων των θεσμικών οργάνων που είχαν λόγο ή που έχουν λόγο, περιλαμβανομένης και της Εποπτικής Επιτροπής της Όλαφ. Τώρα ανακοινώνεται συνεδρίαση με συζήτηση για το αν η ρύθμιση αυτή η οποία έχει ολοκληρωθεί στον τριμερή διάλογο θα ξαναρχίσει διαπραγμάτευση που λέει ότι δεν θα πρέπει να κάνουμε ακριβώς αυτό. Διότι τότε χάνουμε όλες τις επιτευθύνσεις πρόοδους. Τώρα προχωρεί αυτό και έχουμε την υπόθεση Νταλή. Μια υπόθεση που είναι ασφαλώς δύσκολη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου όμως την Επιτροπή αυτή διεξάγεται συζήτηση για το αν η Όλαφ κάνει σωστά τη δουλειά της ή όχι, όπου στην παρούσα Επιτροπή γίνεται συζήτηση για το εάν είναι σωστή η μεταχείριση του κυρίου Νταλή ή όχι. Αυτά θα πρέπει να τα κρίνουν οι δικαστέ στη Μάλτα, όχι εμείς, όχι η παρούσα επιτροπή. Και αυτό είναι σημαντικό να το πει κανείς, διότι δεν έχει και άλλο νόημα αυτή η διαδικασία. Γιατί αυτή τη στιγμή έχει λάβει τη θέση της υπόθεση Νταλή και πολλά που έχουν χρεωθεί στην Όλαφ δεν έχουν αποδειχθεί, συζητούμε για το αν θα ανοίξουμε ξανά το θέμα του κανονισμού της Όλαφ. Εάν η Supervisory, Committee δεν είχε για χρόνια τη δυνατότητα να πει την άποψή της για τον κανονισμό της Όλαφ, Μα υποβάλλεται σήμερα γνωμοδότηση που δεν έχει συνταχθεί, που η συζήτησή της δεν έχει προπαρασκευαστεί και η οποία δεν προκύπτει σαφώς από τα έγγραφα. Και μετά, αγαπητέ Herbert Bush, έρχεσαι και μου λες πράγματα από μια έκθεση που δεν έχει συνταχθεί. Τι είναι αυτή η κομμωδία. Και σε αυτές τις προτάσεις σου ξαναβλέπω πράγματα τα οποία ακούω από την κριτική κατά της Όλαφ στην υπόθεση Νταλή. Αυτά μου φαίνονται πολύ παράξενα. Δεν μιλώ εξ ονόματος ομάδα εργασίας μου και γνωρίζω και μπορώ να διαπιστώσω μάλλον το εξή ότι έχω την μεγάλη ανησυχία ότι αυτή η υπόθεση θα χρησιμοποιηθεί ως δούριος ύπος για να ξαναγίνει μια συζήτηση που εμένα με ενισχύει πάρα πολύ και αρνούμε να συμμετάσχω. Ο Προεδρεύων, ρωτώ τους άλλους και τις άλλες συναδέλφους αν επιθυμεί κάποιος να λάβει το λόγο. Ο κύριος Στάς. Ναι. Με εκπλήσει λίγο η ε, αντίδραση του Γιάννη Γκάιερ, πρέπει να πω. Εγώ τι διαπιστώνω. Το Σάββατο που μας πέρασε κλείνει ε, έξι μήνες από τότε που υποχρεώθηκε να παραιτηθεί ο κύριος Ντάλι. Και θέλω εγώ να δω τι γίνεται. Πριν από 1,5 μήνα ήρθε μια έκθεση από την αποπτική αυτή επιτροπή για τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η έρευνα. Γιατί το ζητήσαμε εμείς αυτό, διότι ακούμε ότι από ό,τι φαίνεται έχουν πάει κάποια πράγματα στραβά στο εσωτερικό της Όλαφ. Και μετά από μεγάλη πίεση ήρθε και η έκθεση της Όλαφ κάπου στο Κοινοβούλιο και η έκθεση της Εποπτικής Επιτροπής είναι απόρριτη αυτή η έκθεση, κάπου την έχουν κλεισμένη σε ένα ντουλάπι, κλειδωμένη και τώρα εμείς θα πρέπει να δώσουμε τις ευλογίες μας για τον νέο κανονισμό που για τα επόμενα 5, 6, 7, 8, 9, 10 πόσα χρόνια ε, θα ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της Όλαφ ενώ γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν προβλήματα ή κάποιες τρευλές πρακτικές. Και πραγματικά με εκπλήσει αυτό που ακούω από τον κύριο Μπεσ. Αν ισχύουν όλα αυτά, θα πρέπει να ανησυχούμε νομίζω εμείς ως νομοθέτες. Και δεν καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά και την αντίδραση του Γιάννη Γκάιερ, ότι δεν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτά τα πράγματα. Τι θα κάνουμε εμείς, πώς θα νομοθετήσουμε για κάτι το οποίο θα ισχύει τα επόμενα δέκα έτη, αλλά ξέρουμε ότι αυτό δρομολογείται με τρόπο που θα είναι δύσκολο να αλλάξουμε το παραμικρό την επόμενη δεκαετία. Ανησυχώ και νομίζω ότι είναι εύλογο να ανησυχούμε. Και δεν κατανοώ και την ηγεσία του Κοινοβουλίου. Διάσκεψη των Προέδρων. Τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου τον ίδιο. Που από ό,τι φαίνεται δεν επιθυμούν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού που είναι στο κάτω-κάτω υπεύθυνα και αρμόδια κατεξοχήν για τον κανονισμό της Όλαφ να μην βλέπουν σημαντικά έγγραφα. Με αυτή η ιστορία με τη Eurostat, το σκάνδαλο του 2002-2003, το θυμάστε? Και ε, έφτασε και στο 10 αυτή η υπόθεση. Διάβασα την απόφαση, τη μελέτησα προσεκτικά και στο σκάνδαλο της Eurostat ήταν δύο ε, υποθέσεις στη Γαλλία και στο Λουξεμβούργο οι έρευνες και παρόλα αυτά ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού είχαμε πρόσβαση και ήμουν και τότε μέλος εγώ και είδαμε τα έγγραφα της Όλαφ, μάλιστα συμμετείχαμε και ε, στη συνεδρίαση ε, της διάσκεψης των Προέδρων των πολιτικών ομάδων πήγαμε τα μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών, ελέγχου μάλλον, για να εξετάσουμε τον Πρόεδρο ε, της Επιτροπής και τον τότε επικεφαλή τον Διευθυντή της Όλαφ και τώρα ξαφνικά τίποτα. Και οποίο διαβάσει την απόφαση του δικαστηριού θα διαπιστώσει ότι... Δεν ε, βασίστηκε η τελική απόφαση του δικαστηρίου σε αυτά τα γεγονότα. Χαίρομαι λοιπόν που τώρα το Εποπτικό Συμβούλιο Επιτροπή αναλαμβάνει τις ευθύνες της. Ήρθανε με ένα προϊόν που δεν έχει ακόμα τελειώσει η έκθεσή τους, μας προειδοποιούν κιόλα, αλλά για μένα τι λέει αυτό, ότι σήμερα σε ό,τι αφορά τον κανονισμό η κατάσταση πραγμάτων είναι τέτοια που δεν μπορούμε να εγκρίνουμε τον κανονισμό. Χρειαζόμαστε περισσότερη πληροφόρηση και ως Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού θα πρέπει να επιμείνουμε και να ζητήσουμε πρόσβαση στα έγγραφα. Από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου το ίδιο. Αλλιώς δεν μπορούμε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Ο πρόεδρος, ο κύριος παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ. Όλα αυτά που ακούω δεν είναι πολύ καθυστυχαστικά. Νομίζω ότι σε αυτή την περιοχή, ε, σε αυτή την επιτροπή, όσο γίνεται πιο σύντομα, πιο γρήγορα να κάνουμε μία συζήτηση για την Όλαφ και όταν τελειώσει και η έκθεση να τη συζητήσουμε, να έρθει ο Διευθυντής της Όλαφ, να, τον, να του υποβάλουμε ερωτήματα, να πούμε ποιες είναι οι περαιτέρω δράσεις που πρέπει να αναλυθούν. Ε, βεβαίως ο καθένας έχει δικαίωμα να απαντήσει σε ε, υποψίες ή κατηγορίες οι οποίες αφορούν το πρόσωπό του και μαζί με τον κύριο Στάς ε, είμαστε από το παλιό αίμα της ε, Επιτροπής αυτής ε, και ίσως και ο πρόεδρος της Επιτροπής μας θα μπορούσε να αποστείλει επιστολή στον διευθυντή της Όλαφ να έχει πρόσβαση στα έγγραφα. Γιατί είχαμε πρόσβαση στην υπόθεση της Eurostat και όχι στην υπόθεση της κυρία, κυρία Λυπάμαι που ξαναζητώ το λόγο, αλλά ο συνάδελφος Γκάιερ ε, χρειάζεται να δεχτεί μια απάντηση. Κοιτάξτε, εδώ δεν πρόκειται για τον Τάλι. Πρόκειται για τον τρόπο με τον οποίο για τις έρευνες για την υπόθεση Ντάλι Όλαφ. Και υπάρχει και ένα όργανο που εμεί το έχουμε ορίσει για να τα ελέγχει όλα αυτά και είναι το Υποπτικό Συμβούλιο, Επιτροπή. Δεν είναι άλλη μια φωνή. Όχι, είναι ε, ο κατεξοχήν αρμόδιος, εμείς τον ορίσαμε για να ε, μα ενημερώνει. Ας μην υποδιόμαστε ότι ήρθε ένα χάρπα στο όργανο τώρα και λέει την αυθαίρετη άποψή του. Εγώ είμαι διατεθειμένη να λάβω αυτή την άποψη πολύ πιο σοβαρά υπόψη από ορισμένους. Τρία θεσμικά όργανα, Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Επιτροπή, έλαβαν την έκθεση της Εποπτικής Επιτροπής τέλη Ιανουαρίου. Ουδής αντέδρασε. Παρόλο που οι παρανομίες ε, ήταν σαφείς εκεί, σύμφωνα με αυτό που μας είπε ο κύριος Μπέρσου. Μα τι Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που δεν εμπιστεύεται στον εαυτό της, δεν τολμάει να καταπολεμά τα κακό κείμενα. Γιατί δεν έχουμε πρόσβαση σε αυτή τη διαδικασία. Και η παραπομπή στη δικαστική, ε, ας πούμε, ε, εξουσία στη Μάλτα είναι ε, παρελκυστική και παραπλανητική και τη δουλειά. Τα πράγματα θα πρέπει να τα έχουμε επιτάπητος, αλλιώς θα έχει αυτό το πράγμα συνέπειες. Δεν μπορούμε να αφήνουμε ένα ευρωπαϊκό όργανο να κάνει πράγματα που δεν επιτρέπονται. Δεν έχουν χειραγωγήσει ολόκληρη έρευνα. Χειραγώγηση είναι αυτό. Ε, δεν το θεωρώ σωστό. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Βγαίνουμε δεξιά και αριστερά και κάνουμε μαθήματα σε όλους και δεν κοιτάμε τι κάνουμε εμείς οι ίδιοι. Α, θα ήθελα να πω και το εξή. Αυτός ο γενικός διευθυντής πρέπει να πούμε ότι είναι πραγματικά αξιοσημείωτα. Χθε κάναμε με τον Μπάρτ κάποιε τροπολογίε και πήρατε όλη ε, ε, αλληλογραφία από την Όλαφ. Αν κοιτάξετε τι λένε εκεί. Εμεί ρωτήσαμε για ποιο λόγο ο Γενικός Διευθυντής κάνει έρευνε. Αυτό ήταν αντικείμενο των δικών μας τροπολογιών. Και λυπάμαι πάρα πολύ ως εισηγήτρια γιατί έχω καταβάλει μεγάλο κόπο ε, για όλο τον κανονισμό. Και με μια τέτοια συμπεριφορά από κάποιον που κάνει οτιδήποτε δεν απαγορεύεται ρητά, το κάνει. Και σε αυτόν τον κανονισμό λίγα πράγματα απαγορεύονται. Λοιπόν, άρα δηλαδή ότι δεν απαγορεύεται επιτρέπεται. Ε, δεν γίνεται αυτό παιδιά. Είναι περίεργη αυτή η κατάσταση και το οικοδόμημα το ευρωπαϊκό περίπλοκο και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Δικαιούται ο Γενικός Διευθυντής να κάνει μόνο του έρευνες νεϊού. Είπε ο κύριο Μπέσο ότι αν το κάνει έχουμε τεράστιο πρόβλημα και αυτό προσπαθήσαμε χτε με τον Μπάρτ να καταδείξουμε. Γιατί βέβαια ο κανονισμό για την Όλαφ του δίνει μια γενική αρμοδιότητα και ευθύνη. Βεβαίω ότι είναι υπεύθυνο για όλου, αλλά δεν είναι και ερευνητή ο ίδιο ο Γενικό Διευθυντή. Θα πρέπει να παραμένει ουδέτερο. Γιατί ακριβώ είναι αρμόδιο και υπεύθυνο για όλα. Δεν μπορεί να κατεβαίνει να κάνει την έρευνα ο ίδιο. Για φανταστείτε. Α μπούμε στο πετσί ενό Ευρωπαίου υπαλλήλου. Τι κάνει ο κακομύρης αυτός. Ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης τον υποχρεώνει να συνεργάζεται με την Όλαφ και να καταθέτει μαρτυρία. Αλλά δεν έχει καμία δυνατότητα να αμυνθεί αν υπάρξει κανένα πρόβλημα παρά μόνο να απευθυνθεί στο ΔΕΚ και θα δικαιωθεί μετά από 10 χρόνια και αν. Από το 2008 η Όλαφ δεν έχει χάσει καμία υπόθεση στο δικαστήριο για παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων. Μα κοιτάξτε πόσο διαρκεί η δικαιοσύνη. Θα δούμε. Ε, ας περιμένουμε. Η απάντηση που μας έστειλε η Όλαφ για μένα είναι πραγματικά χειραγώγηση το κοίταξα και τι να κάνω, μόνο μηδίαμα μου προκαλεί, γιατί τα πράγματα είναι περίπλοκα και όποιος δεν ασχολείται με αυτά τα πράγματα δυσκολεύει. Λοιπόν, είναι χειραγώγηση αυτό και σκάνδαλο το και θα πρέπει και εμείς ξεκάθαρα να λάβουμε θέση. Γι' αυτό ε, ορίσαμε και την εποπτική αυτή επιτροπή για να εποπτεύει, να βλέπει αυτά τα έγγραφα και να το κάνει θέμα. Μα άμα δεν βρούμε εμείς όταν αυτά τα πράγματα βγαίνουν στην επιφάνεια, ε, μπορούμε να το διαλύσουμε το όργανο αυτό, την Εποπτική Επιτροπή, ακόμα και την όλα αυτή ήδη. Γιατί δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έχω κάνει και ερωτήσει στον συνάδελφο Μπέρς και θα ήθελα να μου τις απαντήσει. Όσο γίνεται να έχουμε ευρύτερη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι έρευνες. Όταν κάνουμε τροπολογίες και υπάρχει και λόγος να τις υποβάλουμε, να κάνουμε τις σωστές τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω άλλη παρέμβαση. Άρα παρακαλώ τον κύριο Μπεσ να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για την πρώτη ερώτηση της εισηγήτριας δεν μπορώ να κρίνω παραπέρα. Για τη δεύτερη ερώτηση, εάν πιστεύουμε ότι κάποια θεμελιώδη δικαιώματα θίγονται, εγώ θεωρώ ότι ναι, όντως η απάντηση είναι καταφατική. Να απαντήσω κάτι σχετικά με την ερμηνεία που δίνουμε. Νομίζω ότι οφείλουμε στο Κοινοβούλιο όταν βρισκόμαστε ακριβώς πριν από την έκδοση ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων της Όλαφ, έχει δίκιο η συγκεκριά, αυτή είναι η δουλειά μας, είναι το καθήκον μας. Αυτό μας ανέθεσαν τα τρία θεσμικά όργανα, Συμβούλιο, Κοινοβούλιο και Επιτροπή. Όταν βρισκόμαστε λοιπόν ακριβώς πριν από την έκδοση τέτοια εκθέσεως, εμείς λοιπόν το θεωρούμε ως καθήκον μας να ενημερώσουμε το Κοινοβούλιο και τον Επίτροπο ΣΕΜΕΤΑ άλλωστε για την επικείμενη εκδοσή της εκθέσεως και, το working, και του Working Document, του εγγράφου εργασίας, να ενημερώσουμε, επαναλαμβάνω, το Κοινοβούλιο, διότι θα ήταν αφόρητο, κατά τη γνώμη μου, εάν μπορούσε να μας μεμφθεί το Κοινοβούλιο ότι προχωρήσαμε εμείς, δηλαδή το Κοινοβούλιο, με την ψήφιση αυτής της μεταρρύθμισης και εσείς γνωρίζοντας ότι υπάρχει αυτή η εξέλιξη δεν μας ενημερώσατε. Αυτό θα ήταν λάθος. Και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι δικαιολογημένο, επανέρχομαι, και από σεβασμό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο μας συνδιόρισε μαζί με τα άλλα όργανα, να ενημερώσουμε σήμερα, όπως σήμερα, που ίσως η ενημέρωση αυτή να μην είναι απόλυτα λεπτομερής. Το τι θα κάνει την ενημέρωση αυτή βεβαίως είναι υπόθεση του σώματός σας. για το πότε θα μπορέσουμε να εκδώσουμε την ετήσια, την εγκρίνουμε μάλλον την ετήσια έκθεση, νομίζω θα είναι περίπου 14 με 15 Απριλίου η επόμενη συνεδρίασή μας δηλαδή. Και τότε ασφαλώς θα διαβιβάσουμε το κείμενο στα όργανα εκείνα τα οποία μας ανέθεσαν το εποπτικό έργο. Και νομίζω ότι αυτή είναι σωστή αντίληψη των καθηκόντων μας. Και ευχαριστώ θα σας ευχαριστήσω ιδιαίτερος εάν η ερμηνεία μας αυτή βρει κατανόηση εδώ μεταξύ ημών. Σας ευχαριστώ κύριε Μπες, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι. Εδώ κλείνει αυτό το σημείο της ημερησίας διατάξεως που είναι το πρώτο τελευταίο και μένει το τελευταίο τροποποίηση του κανονισμού 1073 κάθετος 99 σχετικά με έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης Απατών όπου η συγγήτρια είναι η κυρία Γκρέσλε, έχετε το λόγο. Βεβαίως, το θέμα αυτό συνδέεται άμεσα με τα όσα μόλις ακούσαμε. Γι' αυτό και ζήτησα παράταση προθεσμίας. Το Συμβούλιο τα πέρασε τα αποτελέσματα αυτά. Εγώ το θεωρώ και αναγκαίο στο φως αυτών των συμπερασμάτων και που έχουν περιληφθεί σε αυτήν την δυστυχώς μη προσβάσιμη για μας έκθεση για να έχουμε την βάση δηλαδή για τροπολογίες προβλέπεται ωστόσο στους διαδικαστικούς κανόνες η δυνατότητα αυτή. Όταν δηλαδή σημειώνονται νέες εξελίξεις που, ότι, που, που νομίζω ότι συμβαίνει εδώ, μπορούν να κατατεθούν τροπολογίες. Εγώ βεβαίως δεν γνωρίζω προς ποια κατεύθυνση, διότι για να το γνωρίζω θα έπρεπε να μπορέσω να αναγνώσω τα έγγραφα. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να μας δοθούν τα έγγραφα. Για την ώρα έχουμε ζητήσει παράταση προθεσμίας και ελπίζω ότι θα δοθεί αυτή η παράταση. Κατά τα άλλα, το μόνο που μπορώ να πράξω είναι να συστήσω να μην εγκριθεί το κείμενο του κανονισμού. Ως έχει. Ευχαριστώ κυρία Κρέσλε, λέει ο πρόεδρος κύριος Ντόιτς. Έχετε ερωτήσεις ή σχόλια. Επιθυμεί κανείς να λάβει το λόγο. Κυρία Κρέσλε, σας ερωτώ αυτά που είπατε σημαίνουν ότι εδώ οφείλουμε να λάβουμε κάποια απόφαση ή απλώς ήταν ενημερωτικού χαρακτήρα η παρέμβασή σας και επομένως συνεχίζεται η πορεία. Βλέπω ότι νεύεται καταφατικά. Επομένως η απάντηση σας είναι ναι. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή κανείς άλλος δεν επιθυμεί να λάβει τον λόγο. Α, με συγχωρείτε εσείς. Εσείς από άποψη διαδικασίας έπρεπε το θέμα να εγγραφεί σήμερα διότι το Συμβούλιο έχει εγκρίνει το σχέδιο. Υπήρχε λοιπόν από χρόνο λόγος να συζητηθεί σήμερα και θα ήταν σωστό και η σοσιαλιστική ομάδα να αντιληφθεί τη σημασία του αποχρόντος αυτού λόγου. ο Προεδρεύων. Θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Όλαφ. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου κύριε Πρόεδρε να ομιλήσω εξ ονόματος της Επιτροπής και της Όλαφ και να πω λίγα λόγια διότι το θέμα του κανονισμού της Όλαφ βεβαίως έχει εγγραφεί στην ημερησία διαταξή σας. Θα ήθελα πρώτα από άψη τυπική να πω ότι το Συμβούλιο έχει εγκρίνει την θέση του στις 25 Φεβρουαρίου και η Κομισιόν ενέκρινε, το Συλλογικό Σώμα των Επιτρόπων δηλαδή, θέση η οποία υποστηρίζει τη θέση του Συμβουλίου. Επ' αυτού επισημαίνω, όπως άλλωστε είπε και η κυρία Κρέσλε, ότι πάνω από ένα χρόνο σε τριμερείς διαλόγους υπό την διεύθυνση της συζητήσεως της κυρίας Γκρέσλε έγινε η εκπόνηση του κανονισμού της Όλαφ. Και νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι όντως καταλήξατε σε ορθό συμβιβασμό. Η Κομισιόν για την οποία, εξωτερικό της οποίας ομιλώ σήμερα θα θεωρούσε κρίμα και δυστυχές ή ατυχές εάν ο κανονισμός της Όλαφ καθυστερήσει λόγω της καταθέσεως τροπολογιών. Ο κύριος Τόιρερ, επικεφαλής της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, τον Οκτώβριο του 2012 έγραψε επιστολή στην τότε Προεδρία που έδινε πολιτική στήριξη στα πορίσματα του τριμερούς διαλόγου. Επίσης επισημαίνω ότι η ίδια η πρόταση χρονολογείται από το 2006. Έχουν σχεδόν περάσει 7 έτη. Εάν τώρα κατατεθούν ουσιώδει τροπολογίες, όπως ασφαλώς έχει το δικαίωμα το Κοινοβουλίο, δεν αμφισβητώ το δικαίωμα αυτό, είναι αυτονόητο, θα καταστεί όμως δυσχερές να εγκριθεί το κείμενο μέσα στην παρούσα θητεία. Άρα θα χρειαστεί να ανοίξει ξανά νέο κεφάλαιο. Απευθύνω έκκληση λοιπόν και στους βουλευτές της Επιτροπής Ελέγχου Προπολισμού να δείτε το αποτέλεσμα αυτό ως ένα συνολικό θετικό αποτέλεσμα και νομίζω και σε ό,τι αφορά την Εποπτική Επιτροπή η Κομισιόν θεωρεί ότι έχουμε, ε, πρέπει να υπάρχει μια ε, εποπτική επιτροπή της οποίας τα καθήκοντα θα περιγράφονται καλύτερα από ό,τι στον παρόντα κανονισμό. Έτσι, στην πρόταση κανονισμού, βεβαίω μπορεί να πείτε ότι έχουν ε, σημειωθεί κάποιες ανομαλίες. Ο Γενικός Διευθυντής απάντησε στις σχετικές κριτικές. Επί της ουσίας βρισκόμαστε σε διάλογο με την Εποπτική Επιτροπή αλλά αυτό για την ώρα κινείται μεταξύ Όλαφ και Εποπτικής Επιτροπής. Πρόκειται μια ιδιαίτερη υπόθεση η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό συζήτηση και η οποία δεν θα έπρεπε να χρησιμεύσει, να αφορμή για να ανασταλεί η πορεία του κανονισμού. Αυτή είναι η θέση της Κομισιόν και θα ήμουν ευγνώμων εάν είναι δυνατόν να δεχτείτε θετικά αυτήν την ένστασή μου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Επειδή απίθυνε η κυρία Γκρέσλε έκκληση στους σοσιαλιστές να λάβουν υπόψη το θέμα, μπορούμε όντως να το πράξουμε. Έχουν, όπως είπατε, σημειωθεί κάποιες ανομαλίες. Κατανοούμε κάποια απογοήτευση, ότι υπάρχει κάποια απογοήτευση της ε, συναδέλφου μας κυρίας Γκρέσλε, που είναι πράγματι κρίμα γιατί έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά. Εγώ ήμουν σκιώδης συγητής και όντως πρόκειται για ειδικό έγγραφο το οποίο απαιτεί ειδικέ γνώσεις και δεν είναι προσβάσιμο σε όλους, σε ορισμένους τομείς, και να μην είναι απαραίτητο δεκάδες ανθρώπων να κατανοούν το κείμενο αυτό ή να ερμηνεύουν το κείμενο αυτό με τον ίδιο τρόπο της διατάξεις δηλαδή του κανονισμού. Γι' αυτό κατανοώ αυτά που λέει εκπρόσωπος της Επιτροπής ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έστω και αν υπάρχουν διαδικαστικές ανομαλίες δεν θα πρέπει βέβαια να τις παραγνωρίσουμε εργαστήκαμε επί ενός κειμένου επί μια το οποίο ίσως δεν ήταν απόλυτα προσαρμοσμένο. Ίσως και το επόμενο κείμενο να μην είναι τέλειο. Ίσως η ίδια η πραγματικότητα μετά να υπαγορεύσει κάποιες αλλαγές. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να επιδιώξουμε κάποιο συμβιβασμό. Όπως είπα, έχει καταβληθεί σημαντική προσπάθεια και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε εντός της θητείας με τη λήψη μιας απόφασης η οποία ίσως να μην είναι τέλεια αλλά θα είναι όμως δυνατό, θα είναι εφικτή. Παρακαλώ, η κυρία Γκρέσλε. Δεν έχει μικρόφωνο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπέος είναι ακόμη παρόν. Είπε ότι δεν θα πρέπει να λάβει κανείς μια υπόθεση Ω αφορμή για να τρεψει όλο το κείμενο. Αλλά ο κ. Μπέσ είπε ότι είναι μία υπόθεση, αλλά στην πραγματικότητα είναι μία ή πολλέ υποθέσει όπου έχουν γίνει και παρακολουθήσει και μαγνητοφωνήσει τηλεφωνημάτων κλπ. Και δεν είναι απλή υπόθεση μια μαγνητοφώνηση τηλεφωνήματος. Εγώ θεωρώ ότι είναι βαρύνουσα περίπτωση. Λοιπόν, είναι μία περίπτωση μόνο ή είναι πλείονες. Είναι συστημικό το πρόβλημα. Εγώ έτσι κατενόησα ότι πρόκειται για συστημικό πρόβλημα. Και επειδή είναι τέτοιο, νομίζω ότι ο κανονισμός πρέπει να τα διευκρινίζει τα πράγματα αυτά, που δεν το πράττει. Μέχρι τώρα μας φαινόταν εξωπραγματικό ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Γι' αυτό ερώτηση προς τον κύριο Μπέσ και την κυρία Χόφμαν. Ας μου απαντήσουν. Ο Πρόεδρος, η ε, κυρία Χόφμαν, ο κύριος Μπέρς επιθυμούν να απαντήσουν στην ερώτηση αυτή. Ο κύριος Μπέρς πρώτος. Παρόλο που προηγούνται οι κυρίες συνήθως, τώρα είναι λίγο αγενές αυτός. Ο κύριος Μπέρς. Η πρόθεση μας δεν είναι στην αιτήση αυτή η έκθεση να ασχοληθούμε με μεμονωμένες περιπτώσεις ναι. ε, ε, δίνουμε μια εποπτεία για μια επισκόπηση. Είναι πολλές οι περιπτώσεις που μας έχουν απασχολήσει. Καμιά φορά αυτό τι είναι να λησμονείται. Ε, είναι αρκετά σοβαρό αυτό όταν το διαπιστώνουμε και λέγουμε ότι ε, θίγονται κατά την άποψή μας θεμελιώδη δικαιώματα και έχουν θυγεί από έρευνες της υπηρεσίας καταπολέμησης απάτης. Και αυτά τα λέγουμε και θέλουμε να τα διαβιβάσουμε σε εκείνους που φέρουν τελικά την πολιτική ευθύνη για το μέλλον της Όλαφ, έτσι δεν είναι. Ευχαριστώ, κυρία Χόφμαν. Καλά, δεν τρέχει και τίποτα να μιλήσει πρώτος ο κύριος Μπέος. Είμαστε υπέρ της ισότητας, μπορεί να ε, προηγείται και ένας άνδρας καμιά φορά. Λοιπόν, επί της ουσίας νομίζω δεν έχει νόημα να μπούμε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις για να συζητήσουμε για μια συγκεκριμένη έρευνα που μπορεί να δίστανται και οι απόψεις ε, για τα βήματα και τα μέτρα που ακολουθεί και η Όλαφ και η Υποπτική Επιτροπή. Εγώ δεν συμμετέχω τώρα σε καμία έρευνα και δεν μπορώ να αποφανθώ επί του θέματος. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είναι προφανές ότι η γνωμοδότηση της Εποπτικής Επιτροπής απευθύνεται και σε Όλαφ, Αν το δείτε και στον κανονισμό το λέει αυτό. Και βεβαίως θα τη μελετήσουμε πάρα πολύ προσεκτικά. Απαντήσαμε ε, και η Όλαφ και ο κύριος Κέσλερ, ο Γενικός Διευθυντής και οι συνάδελφοι είναι πάντα πρόθυμοι να το συζητούν αυτό επί της ουσίας με την Εποπτική Επιτροπή. Μπορεί να μην συμφωνούμε πάντα με την Εποπτική Επιτροπή σε όλα τα θέματα, μα γι' αυτό υπάρχει άλλωστε για να συνεννοούμαστε, να συζητούμε και είμαστε πρόθυμοι πάντα να το κάνουμε. Ο κύριος Κέσλερ δεν έχει κανένα πρόβλημα, ο γενικός μας διευθυντής να έρθει στην Επιτροπή σας να αναφέρει και πάλι. Ε, νομίζω είναι πολύ μεγάλη διαφάνεια εδώ. Ε, ε, κατά την άποψή μας λοιπόν, δεν έχουμε ε, παραβιάσει σε καμία περίπτωση σοβαρά το δικαίωμα και αυτό το αποκρούω ε, πραγματικά ε, με επιμονή. Μπορεί να υπάρχουν κάποια ζητήματα, αλλά δεν δικαιολογεί αυτό να αναβάλλεται μια νομοθεσία που δεν έχει καμία άμεση σχέση με την λόγω υπόθεση. Η κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι. Λυπάμαι που δεν μπόρεσα να είμαι παρούσα για να ακούσω τα όσα είπε ο κύριος Μπέρς, γιατί είχαμε άλλο πρόβλημα στην Επιτροπή Μεταφορών. Θα ήθελα όμως να σχολιάσω κάτι, να πω στην κυρία Χόφμαν και να τη θυμίσω ότι όταν για πρώτη φορά ε, ε, συναντηθήκαμε με τον κύριο Κέσλε, δημόσια στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού με τον Γενικό Διευθυντή της Όλαφ, υπήρξε μια πρώτη αντίδραση Γιατί έλεγε ο κύριος Κέσλερ ότι η Εποπτική Επιτροπή δεν χρειαζόταν να έχει ε, όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες που ήθελε να τις δώσει το Κοινοβούλιο. Δηλαδή ήδη από τότε υπήρχε κάποια επιφύλαξη. Μιλάτε για μία υπόθεση, δεν είναι οποιαδήποτε υπόθεση, είναι μία υπόθεση ε, ε, που αφορά την εκτελεστική εξουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει εμπλακεί σε μία κατάσταση έτσι κάπως τραγελαφική ε, και είναι και ένα νομοθέτημα πάρα πολύ σημαντικό ε, αφορούσε και τον καπνό ξέρετε αυτές τις ιστορίες ήταν και σε πλήρη προεκλογική εκστρατεία ε, και ο ε, λόγω ο κύριος που υποχρεώθηκε σε παρέτηση προσφεύγει τώρα. Ε, εντάξει, το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να διευκρινιστεί τουλάχιστον αυτή η υπόθεση, γιατί το απαιτούν και οι Ευρωπαίοι πολίτες. Δεν μπορούμε να μιλούμε μόνο για ε, απλές διοικητικές δυσλειτουργίες παραβλέψεις ή σφάλματα. Δεν είναι η πρώτη φορά που καταδικάζεται η Όλαφ για υπέρβαση καθήκοντος και αρμοδιοτήτων και μάλιστα κατόπιν εορτής. Άμα περάσουν και τόσα χρόνια είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποκατασταθεί η τιμή κάποιων ανθρώπων, η περιουσία τους κτλ. Και υπήρχαν και ίσονος σημασία υποθέσεις. Ο κύριος Ντάλι όμως δεν είναι άλλη μία υπόθεση, είναι η υπόθεση. Το είπε και ο κύριος Βαλτσίτης και η κυρία Γκρέσλε. Ε, η κυρία Γκλέσσα που έχει κάνει όλη αυτή τη δουλειά, αν μας ζητάει να βελτιώσουμε ε, την κατάσταση δεδομένη της τελευταίας υπόθεσης που επαναλαμβάνω δεν είναι μια τυχαία υπόθεση γιατί έχουν προκύψει νέα στοιχεία λοιπόν ας μελετήσουμε τα στοιχεία αυτά και τέλος θα ήθελα επίσης να ρωτήσω κάτι απλώς δεν ξέρω ποιος θα μου απαντήσει αν μπορεί η κυρία Χόφμα να μας απαντήσει γιατί και πάλι είναι θέμα περιπτωσιολογίας. Τι θα συμβεί λοιπόν σε περίπτωση που το δικαστήριο στη Μάλτα θεωρήσει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Δικαιώσει τον κύριο Ντάλι λοιπόν. Τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Υπάρχουν συνέπειες. Τι θα γίνει λοιπόν ε, εάν αθωθεί από το δικαστήριο στη Μάλτα. Ε, ο πρόεδρο. έκανε μια ερώτηση κυρία Γιάλα. Δεν θέλω να περιορίσω κανέναν στην έκφραση ε, της άποψής τους, ε, αλλά κατά την άποψή μου δεν είναι δική μας δουλειά να ασχοληθούμε επί της ουσίας ε, με μια απόφαση που κρεμεί τη δικαιοσύνη και να προεξοφλήσουμε και να προδικάσουμε και το, την απόφαση του δικαστηρίου και να αναγκάσουμε πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μας απαντήσει γι' αυτό. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να απαντήσει, να σχολιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, αυτό το ερώτημα. Θέλω να δώσω το λόγο στην κυρία Γκρέσλε, αλλά προηγουμένως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Α, επιθυμεί η κυρία Χόφα. Ε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να συνηγορήσω υπέρ αυτού που λέει η Μαργαρίτα Χόφμαν ε, σχετικά ε, με αυτό που θα οφείλαμε να κάνουμε, τι είναι σημαντικό δηλαδή να γίνει ανάμεσα στην ε, υπόθεση που οδήγησε στην παρέτηση του κυρίου Νταλή και υπόθεση για την οποία ε, πρέπει να απαντηθούν και να διευκαλυνθούν πολλά ερωτήματα, όχι απαραίτητα εδώ, αλλά κυρίως ενώπιον των ε, δικαστηρίων και του Ευρωπαϊκού Στείου στο Λουξεμβούργο και ε, του δικαστηρίου στην Μαλτά αφενός και τον κανονισμό Όλαφα Φετέρου. Ο κανονισμός Όλαφα αποτέλεσε αντικείμενο πολλών και εντελεχών συζητήσεων σε όλα τα θεσμικά ε, όργανα και υπήρξε συμφωνία με το Συμβούλιο επ' αυτού το γεγονός ότι ενδεχομένως, γιατί δεν ξέρουμε, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αν υπήρξαν δυσκολίες οι οποίες προκάλεσαν το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης, εάν έχει προκύψει κάποιο πρόβλημα, δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες ε, της έρευνας ε, και δεν έχω την έκθεση. Βεβαίως ε, θα διαβάσουμε με μεγάλη προσοχή και ενδιαφέρον την έκθεση της Εποπτικής Επιτροπής, αλλά αυτό δεν μας αφορά ε, σε σχέση με το γενικότερο κανονισμό. Και εν πάση περιπτώσει, εάν πρέπει να εξαχθούν κάποια συμπεράσματα από μια ειδική περίπτωση, ε, θα πρέπει να το δούμε και να δούμε μήπως ε, ε, μπορεί ο Γενικός Διευθυντής της Όλαφ μέσα από λειτουργικές κατευθυντήριες γραμμές, συγγνώμη επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές να διορθώσει λίγο ή να αποσαφηνίσει κάπως κάποια στοιχεία. Μέχρι τώρα έχουμε και πολύ, μια πολύ καλή διαδρομή και βεβαίως και το Κοινοβούλιο μπορεί να αποφασίσει ενδεχομένως για κάποιες ε, τροπολογίες αλλά κοιτάξτε δεν μπορεί ε, ένας ε, κανονισμός να είναι εξαντλητικός δεν μπορεί να λυθούν όλα στις ελάχιστες λεπτομέρειες σε έναν κανονισμό και ούτε είναι και λογικό άλλωστε Πιστεύω λοιπόν ότι οι επιπτώσεις όλων αυτών των υποθέσεων ή μάλλον τα συμπεράσματα από όλες αυτές τις επισ υποθέσεις, συγγνώμη, θα πρέπει να εξαχθούν. Αλλά πρέπει να πω ότι ο κανονισμός στην παρούσα φάση αναθεώρησης την οποία διανύει αποτελεί μεγάλη πρόοδο σε σχέση με τον αρχικό ε, κανονισμό. Βλέπουμε ότι υπάρχει ενίσχυση δικαιωμάτων στο νέο κανονισμό και επομένως γιατί να καθυστερήσουμε αυτήν την μεγάλη πρόοδο, γιατί να καθυστερήσουμε αυτήν την μεγάλη πρόοδο στις σχέσεις με τις διοικήσεις. Θα ήταν πραγματικά πολύ κρίμα εάν ένα υπομονή των ε, συμπερασμάτων ε, που ίσως ε, πάρουν καιρό μέχρι να εξαχθούν γιατί η δικαιοσύνη είναι λίγο βραδία όπως γνωρίζετε. Γιατί να περιμένουμε λοιπόν ε, και εν πάση περιπτώσει βεβαίως εάν προκύψουν και συγκεκριμένα στοιχεία προφανώς θα ζητηθούν ε, και αποζημιώσεις και αλλά ακόμα δεν βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Έχουμε εδώ έναν ε, κανονισμό αναθεώρηση που είναι σημαντικός και για την Κομισιόν και για την Όλαφ και για τους συμβαλόμενους και για τους εμπλεκόμενους και δεν καταλαβαίνω γιατί μια ειδική περίπτωση πρέπει να μας καθυστερήσει. Δεν είναι λογικό αυτό. Βεβαίως, από την άλλη πλευρά, το να μελετήσουμε προσεκτικά όλες τις εκθέσεις της Εποπτικής Επιτροπής, ε, να εξαχθούν τα απαραίτητα συμπεράσματα, να τα εξάγει και η ίδια η Όλαφ, ε, βεβαίως πρέπει να γίνει αλλά και με την ευκαιρία της έγκρισης του νέου κανονισμού θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε για όλα αυτά. Πιστεύω ότι πρέπει να αποφύγουμε, να καθυστερήσουμε την έγκριση ενός κανονισμού που αποτελεί μεγάλη πρόοδο ε, σε σχέση με ένα κείμενο το οποίο ήδη είναι απαρχαιωμένο γιατί είναι ένα κείμενο του 99. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Πριν κλείσουμε το σημείο αυτό, θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Γκρέσλε, παρακαλώ. Επισημένω και πάλι ότι αυτή η Όλαφ αποτελείται από μεμονωμένες υποθέσεις και ο χειρισμός πολλών επιμέρους υποθέσεων δίνει συνολικά δίνει τελικά την συνολική εικόνα. Η υπόθεση περί την οποία στρέφεται η συζήτηση σήμερα είναι πολύτιμη με την έννοια ότι έχει διερευνηθεί πολύ σε βάθος. Ωστόσο αυτό που βλέπω και εγώ λυπούμε περισσότερο από, καθέ, από καθέναν άλλον που είμαστε υποχρεωμένοι να συζητήσουμε την ιστορία αυτή σήμερα γιατί ήταν τόσο δύσκολο να καταλήξουμε στη συμφωνία γιατί ήταν πραγματικά πολλή δουλειά. Όμως αυτά που αντλούμε από την υπόθεση αυτή, ίσως και από άλλες, είναι Δεν μπορώ να σας δω κυρία Χόφμαν, μου κάνει εντύπωση ο τρόπος με, την, με τον οποίο εμφανίζεστε εδώ. Δεν το βρίσκω σύνηθες, μια πολίτης η οποία τυχαίνει και είναι μέλος λόμπι για προϊόντα καπνού ενθαρρύνεται να μαγνητοφωνήσει τηλεφώνημα. Εγώ όταν μιλώ για έρευνα κατανοώ ότι συλλέγονται οι ενδείξεις και οι αποδείξεις που υπάρχουν ήδη, όχι ότι φτιάχνονται. Κάποια στιγμή θα ξεπηδήσει αυτή η ιστορία. Αλλά αυτό που μου κάνει μεγάλη εντύπωση είναι ότι όλα πρέπει να μπουν σε διατάξεις απαγορεύεται ή επιτρέπεται, γιατί αλλιώς γίνεται οτιδήποτε να απαγορεύεται. Έχω εγώ υποβάλει και γραπτές ερωτήσεις. Η Όλαφ έχει διαβάσει πράγματα και στους συναδέλφους που δείχνει ότι δεν αντιλαμβάνονται καν το πρόβλημα. Αυτό με αφήνει με το στόμα ανοιχτό. Δεν υπάρχει απόλυτα καμιά συνειδητοποίηση των προβλημάτων για αυτό το ε, αβέβαιο νομικό έδαφος στο οποίο κινούνται. Δεν αντέχει αυτό τέτοιου είδους ε, εμφάνιση από την πλευρά των εκπροσώπων της Όλαφ. Δεν μπορεί να εμφανίζεται με τον τρόπο αυτό. Οι αξιωματούχοι της Ένωσης και μεταξύ αυτών των αξιωματούχων έχω μάλλον περιορισμένο αριθμό φίλων. Αυτά που μπορεί ενδεχομένως να κάνει όλα Όλαφ σε βάρος των αξιωματούχων της Ένωσης δεν είναι δυνατόν. Και έρχομαι τώρα στις δάσεις επαιγές Κέμπρη. Μου φαίνεται απίστευτο ο τρόπος με τον οποίο αφαιρέθηκε από την αρχή από την εργασία της Εποπτικής Επιτροπής με χειρισμούς, με χειραγώγηση διαδικασίας. Δεν μπορείτε να μου πλασάρετε τα πράγματα αυτά που έρχεστε και μου λέτε εδώ. Είμαι γνώση των θεμάτων. Δεν μπορείτε να έχετε να μου λέτε τέτοια πράγματα. Ξαναλέω, μένω με το στόμα ανοιχτό απέναντι σε αυτή τη συλλογή μισών αληθιών, ας το πω έτσι. Τα πράγματα αυτά πρέπει να τεθούν επιτάπητος. Εάν όχι, τότε θα μετανοήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται η Όλαφ και η Κομισιόν. Χρειαζόμαστε λοιπόν πλήρη εικόνα της ιστορίας αυτής. Το καλύτερο είναι κάντε το εσείς οι ίδιοι. Αυτό είναι το προτιμότερο. Ε, πραγματικά αισθάνομαι σοκ από τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται ορισμένα πράγματα. Αυτές οι οδηγίες προς το προσωπικό. Εσύ συμμετέσχες στην έκδοση αυτού του εγχειριδίου με τους κανόνες διαδικασίας της Όλαφ. Και εγώ αγωνίστηκα. Ήταν σαφές ότι ήταν πολύ δύσκολο να περάσει από τη συναπόφαση αποδείχνεται τώρα ότι με αυτές τις instructions του staff κάνουν θέλουν. Αν κατάλαβα καλά από τα όσα είπαν οι εκπρόσωποι της Κομισιόν. Εγώ ανέμενα ότι οι instructions του staff θα είναι δεσμευτικές και μεταφράζονται και σε όλες τις γλώσσες μάλλον, είναι δημόσιες. Είναι λοιπόν τμήμα της διαδικασίας και επομένως τμήμα της προστασίας των θεμελιδών δικαιωμάτων. Φαίνεται πως τώρα όμως θεωρούν ότι δεν είναι δεσμευτικέ οι διατάξει αυτέ και μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ το βρίσκω αυτό καταστροφικό. Είναι καθαρά ενάντια στο πνεύμα των όσων διαπραγματευτήκαμε. Κοιτάξτε τώρα. Τι γίνεται, πράγματα που γίνονται δηλαδή που είναι αντίθετα με το πνεύμα της ρύθμισης. Εγώ ευχαρίστως να συμφωνούσα αλλά δεν είναι δυνατόν να κάνετε πράγματα τα οποία είναι σαφές, σαφής παραβίαση του δικαίου. Από α μέχρι το, τελ, μέχρι το, β, μέχρι ω. Έχω την εντύπωση ότι δεν αντιλαμβάνονται καθόλου το τι λέω. Λάβετε το σοβαρά υπόψη σας αυτά. Εγώ λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη τα όσα λέει ο Γενικός Διευθυντής. Και διαρωτώ με, τι σημαίνουν αυτά που λέει, τι σημαίνουν, τι σημαίνουν αυτά που κάνει. Κάντε και εσείς το ίδιο και επανερχόμαστε τότε, επανερχόμαστε και ξανασυζητούμε. Ευχαριστώ κυρίε και κύριοι συνάδελφοι. Εδώ ολοκληρώνεται η συζήτηση αυτού του θέματος της ημερησίας διατάξεως και λάβαμε υπόψη τα όσα δήλωσε η κυρία ε, Γκρέσλε ως εισηγήτρια. Επιθυμείτε να θέσετε θέμα διαδικαστικό. Ε, ναι. Κοιτάξτε κύριε Μπέρκ, δεν ε, ξέρουμε όλες τις λεπτομέρειες της κατάστασης. Ε, συζητάμε την απόφαση εδώ και μισή ώρα, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς περί τι πρόκειται. Έχουμε κάποια στοιχεία ότι κάτι συμβαίνει, έχουμε ακούσει κάποιες φήμες, έχουμε ακούσει κάποια στοιχεία χωρίς να τα έχουμε δει όλα. Δεν νομίζετε ότι είναι δικαιολογημένο το ότι ζητούμε τα ε, έγγραφα. Επισήμως έχουμε ζητήσει τα έγγραφα αυτά. Ε, ίσως θα πρέπει ξανά να τα ζητήσει ο Πρόεδρος της Επιτροπής μας. Όχι για ευρεία δημόσια κυκλοφορία, για τα μέλη της Επιτροπής για να τα έχουμε. Έτσι, να, έτσι ώστε να έχουμε και την απαραίτητη πληροφόρηση γιατί διαφορετικά. Είναι σκανδαλώδες αυτή η κατάσταση. Ε, συζητούμε, ξανασυζητούμε. Λέμε αυτό δεν είναι αλήθεια, είναι ίσως αλήθεια, ενδεχομένως συνέβη, μπορεί ο κανονισμός να εφαρμόζεται και με άλλο τρόπο. Τι να σας πω τώρα, συμφωνώ με την κυρία Γκρέσλε ότι θα πρέπει να αναλύσουμε την περίπτωση αυτή εν λεπτομερία και τότε ίσως τα συμπεράσματά μας να είναι και διαφορετικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βουλευτά. Προσωπικά Ε, πρότεινα να ολοκληρώσουμε εδώ το σημείο αυτό της μέσης δέδαξης, Να ευχαριστήσουμε την κυρία Γκρέσλε και να σημειώσουμε ότι θα απευθυνθώ στον πρόεδρο της Επιτροπής μας για τα θέματα που ανέκυψαν, έτσι ώστε τα ερωτήματα αυτά να απαντηθούν τελικά να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση στα έγγραφα, τα οποία υπάρχουν έτσι και αλλιώς στο Κοινοβούλιο. Λοιπόν, θα ε, κάνω τα απαραίτητα βήματα. Στα διάφορα δεν έχω τίποτα. Έχει κανείς τίποτα να προσθέσει στα διάφορα στο 59, όχι. Ωραία. Σας ευχαριστώ. Προσεχή συνεδρίαση στις 23 Απριλίου 2013 στις 3 το μεσημέρι στις Βρυξέλλες. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Χαίρετε.